Merci. Alors je ne suis pas venu tout seul. Euh, les enfants euh, viennent d'une école qui qui s'appelle. Τα παιδιά έρχονται από ένα δημόσιο σχολείο που λέγεται Λεγκριότ, τα Πετροκέρασα.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

bien, bravo les enfants, hein. Μπράβο στα παιδιά, λέει ο πρόεδρο. Vous chantez beaucoup mieux que moi. Τραγουδάτε σίγουρα καλύτερα από μένα. Μη φοβάστε, δεν θα τραγουδήσω. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τους καθηγητές σας. Αντιπρόεδρε Μογκερίνη, κύριε Κασλέ, είναι τιμή μου που σας καλωσορίζω στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα 70 χρόνια της διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Παρίσι το 48. Η νεόκοπη τότε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το κείμενο αυτό το οποίο προβλέπει ότι το ανθρώπινο όν επειδή υπάρχει έχει δικαιώματα. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο μπορεί να μην είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του αλλά έχει ιστορική και συμβολική σημασία πάνω από 90 χώρες αναφέρονται στα συντάγματά του στο συγκεκριμένο αυτό έγγραφο. Η προστασία όμως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυστυχώς υπόκειται σήμερα νέου τύπου απειλές. νέου τύπου απειλές. Η ελευθερία έκφρασης ε, αντιμετωπίζεται με στρεβλό τρόπο και οδηγεί ε, σε παραβίαση της ε, ιδιωτικότητας, το ίδιο επίσης ε, και η διαχείριση των ψευδεπίγραφων νέων και ειδήσεων, συν της τα δημογραφικά προβλήματα, οι ανθρωπιστικές κρίσεις και οι σειράξεις που χαίνουν στον κόσμο σήμερα οδηγούν σε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό έχει δραματικές συνέπειες για τους πληθυσμούς οδηγούν στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και στην καταστολή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να εμείνουμε στην δήλωση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες και τις αρχές που εμπεριέχει. Οι βασικές αυτές αρχές είναι και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ζήσει τη φρίκη των δύο παγκοσμίων πολέμων και της παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι προσπάθησαν αυτές τις τραγωδίες να μην τις επαναλάβει η Ευρώπη. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και του κράτους δικαίου επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγγυηθεί 70 ολόκληρα χρόνια ειρήνης Όλα αυτά ορίζονται από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκές και εκφράζονται μέσω και της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μοναδικά, μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο, υπερασπίζεται ε, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και 30 χρόνια με το βραβείο Ζαχάροφ από τη φοροτιμή σε πρόσωπα και οργανώσεις που κρατούν ψηλά το λάβαρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέντε νικητές άλλωστε του βραβείου Σαχάροφ πήραν και το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. Και η Εβδομάδα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποδεικνύει θα έλεγα την αφοσίωσή μας. Πρέπει να Ευχαριστήσουμε λοιπόν καθημερινά τις οργανώσεις που δίνουν μάχες καθημερινά ε, για να διασώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη. Πολλές από τις οργανώσεις αυτές είναι παρούσες εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Είστε οι θεματοφύλακες των δικαιωμάτων όλων μας. Σήμερα είναι η μέρα των δικαιωμάτων επίσης ε, της νεαρής ηλικία των παιδιών. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά μεταξύ μας, τα οποία με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση καλωσορίζω. Εκπροσωπούν το μέλλον μας και ελπίζω το μέλλον αυτό και το δικό τους μέλλον να είναι καλύτερο από το παρόν γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις βίας υπάρχει βία εις βάρος των παιδιών, σεξουαλική βία υπάρχουν ε, θύματα πολέμου ε, ανάμεσα στα παιδιά. Πρέπει λοιπόν χωρίς να σταματήσουμε καθόλου να προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε το μέλλον σας. Σε αυτό το μεγάλο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει όλοι να νιώθετε προστατευμένοι και θα πρέπει επίσης να προσπαθείτε να συμμετέχετε και να επηρεάζετε τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Αυτή είναι η δημοκρατία θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά μέσα και το διαδίκτυο χωρίς να αντιμετωπίζετε ε, κινδύνους από αυτά τα οποία ε, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και από το cyberbullying. Ε, υπάρχουν μέσα όπως το YouTube, το Netflix, ε, που πρέπει να λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες έτσι ώστε να απομακρύνονται αμέσως τα κατάλληλα περιεχόμενα και να προστατεύονται τα προσωπικά στοιχεία. Νομίζω ότι και η τελευταία έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγινε δεκτή την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ζητά από τα κράτη-μέλη με μία φωνή να στηρίξουν για μια ακόμη φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτούς που τα προασπίζονται. Πρέπει να επιμείνουμε στη συμφωνία αυτή έτσι ώστε κανείς να μην διώκεται για αυτά που πιστεύει ή για την πίστη του. Ε, η Άζια Μπίμπη στο Πακιστάν όπου υπάρχουν πάρα πολλές θρησκευτικέ μειονότητες που υφίστανται τις συνέπειες της καταστολής στον κόσμο. Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε και τους πρωτοπόρους των δικαιωμάτων μας, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να ενημερώσουν σωστά για να διασώσουμε την ελευθερία μας εμείς η Γκαρουάνα Καλίτσια, η Σόζη είναι οι πιο πρόσφατες περιπτώσεις δημοσιογράφων που έχασαν την ίδια τους τη ζωή για να υπερασπιστούν την ίδια την αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι κρατούμενοι στις τουρκικές φυλακές όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου. Οι σημερινές εκδηλώσεις λοιπόν θα πρέπει να είναι καθρέφτης του ότι σε πολλές χώρες δυστυχώς δεν υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων. Πολλές φορές οι γυναίκες στερούνται τα δικά τους θεμελιώδη δικαιώματα παραμερίζονται στις κοινωνικές εξελίξεις και πέφτουν θύματα της βίας. Ανανεώνω λοιπόν την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ τι χώρε που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη για τη βία ει βάρο των γυναικών. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και τι συμβαίνει στο εσωτερικό του ίδιου μας του σπιτιού. Πολλές γυναίκες χάνουν τη ζωή τους δυστυχώς και πολλές γυναίκες αντιμετωπίζονται με βία. Πολλές γυναίκες θεωρούνται ότι είναι κατώτερα όντα Αυτά συμβαίνουν, μπορεί να συμβούν και εδώ ακόμα. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε επίσης και την κατάσταση σε χώρες όπως τη Βενεζουέλα. και εκεί παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν αυθαίρετες συλλήψεις και φυλακίσεις και παραβιάζεται η ελευθερία έκφρασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα, υποστηρίζει τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, υποστηρίζει τους πρασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή όπως αυτούς οι οποίοι ε, πήραν το βραβείο Σαχάροφ το 2017. Η κυρία Μπασλέ η οποία είναι τέος πρόεδρος στη Χιλή και υπεύθυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως Νότιο-Αμερικάνα έχει προτεραιότητα για να μιλήσει για αυτή την κατάσταση. Κλείνοντας να θυμίσω την Έλενο Ρούσβελτ η οποία έλεγε ότι οι διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις δεν παίζουν ρόλο όταν απλά ο κόσμος τις γνωρίζει, αλλά όταν ο κόσμος, όταν οι πολίτες απαιτούν να παίρνουν ζωή και να εφαρμόζονται. Γιατί δυστυχώς ο κόσμος τον οποίο ζούμε σήμερα περιλαμβάνει και ρητορικές καταστροφικές και λαϊκιστικές και γι' αυτό θα πρέπει ακριβώς αυτό το έγγραφο που μας ενδιαφέρει σήμερα να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να απομακρύνουμε αυτούς που απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ας γίνουμε όλοι πρωταθλητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας ζητήσουμε και από τις κυβερνήσεις και από την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε στις Βρυξέλλες. Να δώσω το λόγο τώρα στην ύπατη εκπρόσωπο, την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη. Μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε μέσω βίντεο το Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτιέρεθ. Grazie Αντώνιο, Ευχαριστώ, Αντώνιο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ειλικρινεί ευχαριστίες προς εσένα, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αποφασίσατε να εορτάσουμε από κοινού αυτή την ημέρα. Θεωρήσαμε ότι ίσως ήταν το καλύτερο να κάνουμε, να διοργανώσουμε εορτασμό για την επέτειο της διακήρυξης της οικουμενικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μαζί με το ετήσιο φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, πιστεύω ότι ήταν ε, έξοχη αυτή η ευκαιρία για να δείξουμε πώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μαζί εργάζονται για να προστατεύσουν και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο σε συνεργασία με του φίλου μα τη κοινωνία των πολιτών. 70 χρόνια μετά τη διακήρυξη των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ετοιμάστηκε η Χάρτα, ακόμα εργαζόμεθα να μετατρέψουμε τα λόγια τη διακήρυξη σε πρακτική. Και ένα μεγάλο τμήμα τη συλλογική εργασία γίνεται από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και ειλικρινέστατα εσάς από τι οργανώσει κοινωνία των πολιτών και εκείνους που εργάζονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φίλου από όλο τον κόσμο, με του οποίου καθημερινά συνεργάζεστε στι χώρε σα και οι οποίοι σήμερα έκανε το ταξίδι για να έρθουν εδώ και να είναι μαζί μας. Εσεί είσαστε το βασικό κομμάτι τη δουλειά που κάνουμε, να προωθήσουμε και να υπασπιστούμε τα και δικαιώματα. Διαβάζοντα τη διακήρυξη, διαφαίνεται σαφώ ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. 70 χρόνια πριν, η διακήρυξη δήλωνε ότι ο καθένα έχει το δικαίωμα στην εργασία και το δικαίωμα σε ίση αμοιβή για ίση εργασία αναγνώρισε όλα τα δικαίωμα όλων στην παιδεία, χωρίς διάκριση αφορά το φύλλο, το γένος, εθνικότητα, θρησκεία, κοινωνικό υπόβαθρο και, τα, και οικονομικούς πόρους. Η διακήρυξη ήταν μπροστά την εποχή της. Στην Ιταλία, στη χώρα μας, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να ψηφίσουν μέχρι μόλι ε, μόλις δύο χρόνια πριν τη διακήρυξη και σε πολλές άλλες χώρες τα δικαιώματα ψήφου ήταν περιορισμένα σε μερικές κοινωνικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά αναγνώρισε η διακήρυξη και παραθέτω ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην ε, διακυβέρνηση της χώρας του και να συμμετέχει στην κυβέρνηση τη χώρας του. Και η βούληση του λαού θα είναι η βάση του κύρου και τη κυριαρχία και τη εξουσία τη κυβερνήσεω. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ούτως ώστε να έχουμε δημοκρατίες που καλύπτουν ομοίωμα όλους και να καλυφθούν οι, οι διαφορές αμοιβών ανάλογα με το φύλλο. Να έχουν όλοι αξιοπρέπεια, να αντιμετωπίζουν αξιοπρέπεια ανεξάρτητα φύλλου, χρώματος και καταγωγής. Όλοι, πολλοί από εσά που είσαστε εδώ αφιερώσετε τη ζωή σας στην εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών και είμαστε γνώμονες γι' αυτό. Και για αυτή την αφοσίωση και προσπάθεια μερικοί από εσά ε, αντιμετωπίσατε φυλάκιση, παρενόχληση, βία Τόσοι πολλοί φίλοι, προσωπικοί σα φίλοι, είναι στη φυλακή. Πολλοί από του συναδέλφου και φίλου δεν μπορούν να παρίστανται εδώ σήμερα μαζί μα, διότι έχασαν την ελευθερία του ή έχασαν τη ζωή του. 70 χρόνια μετά τη διακήρυξη αυτή ε, δεν μπορούμε να θερέσουμε δεδομένα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σήμερα συλλογικά και να περάσει σε όλους μας. Αντίθετα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδει ελευθερίε έχουν δεχτεί νέε πιέσει. Κάποιοι στον κόσμο επιχειρηματολογούν λέγοντα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ξεπερασμένα, απειρχιωμένα, ότι τα εθνικά συμφέροντα μπορούν να δικαιολογήσουν την καταστολή των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, ότι η εθνική ασφάλεια απαιτεί την αναστολή κάποιων δικαιωμάτων. Ε, πιστεύω ότι όλοι είμαστε σήμερα εδώ για να διατρανώσουμε το αντίθετο. Ότι η μόνη βιώσιμη ασφάλεια είναι η ασφάλεια που βασίζεται στο πλήρη σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν τα πολιτικά δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, οι ατομικέ ελευθερίε την χάνουν εγγυήσεων, τότε είναι ισχυρέ πραγματικά και προστατευμένε και ασφαλεί οι κοινωνίε μα. Κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι παραβίαση των συλλογικών και εθνικών συμφερόντων μα. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτου προσπαθήσαμε να το δείξουμε αυτό στην πράξη μέσω πραγματικών ιστοριών ανθρώπων όπω είστε εσεί, παριστάμενοι στην αίθουσα. Σε μια στιγμή που τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση, θέλουμε να μετακινηθούμε από αμυντική προσέγγιση σε μια πιο ε, δραστήρια ε, προσέγγιση, διότι αμφισβητούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να έχουμε υπόψη τι σημαίνει στην πράξη το ανθρώπινο δικαίωμα, στην καθημερινή ζωή και τι έχουμε πετύχει μαζί σε αυτά τα 70 χρόνια από την διακήρυξη των δικαιωμάτων αυτών. Κάποιε από τι χώρε μα δώσαν με το δικαίωμα μελέτη και ψήφου ανθρώπου που δεν το είχαν ποτέ πριν. Εκπαίδευση μάλλον. Και αυτό είναι ισχυρότερο κινητήρα για αλλαγέ. Κάποιε ε, χώρε μα έβγαλαν από τη φτώχεια χιλιάδε ανθρώπου και μπόρεσαν έτσι να συμβάλλουν πληρέστερα στην δημόσια ζωή. Κάποιοι πήγαν από δικτατορίε στη δημοκρατία και στην Ευρώπη ακόμα για να πούμε αυτές τις ιστορίες ενώσαμε τις δυνάμεις με 13 χώρες από όλες τις υπήρους για να δείξουμε ότι η πρόοδος σε αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνει χώρα, πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο και αυτό μόνο χάρη στην αποφασιστικότητά μας και θα έλεγα και στο πείσμα μας και στο θάρρος σας. Και είμαι ευγνώμων προς τον Μισελ διότι είμαστε μαζί στη Νέα Υόρκη κατά τη Γενική Συνέλευση παρουσιάζοντας αυτές τις θετικές καλές ιστορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα δίνοντας η αποφασιστικότητα, το θάρρος και το κοινό έργο δίνει αποτελέσματα. Έχουμε πει, έχουμε διηγηθεί τη ιστορία για να δείξουμε ότι η πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εφικτή και είναι κάτι που συμβαίνει. Χάρη σε ανθρώπου σαν και εσά υπάρχει ελπίδα ότι αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα από σήμερα. Είναι ιστορίε που δίνουν δύναμη, δείχνουν ε, διόρθωση σφαλμάτων, κοινότητε που ισχυροποιούνται, δείχνουν χειραφέτηση, δείχνουν το έργο των διαφόρων οργανώσεων. Τα κορίτσια που αρνήθηκαν παντρευτούν πολύ πρόημα, τη χάνουν ε, βοηθεία και οι ηθαγενείς πληθυσμοί μπορούν να ζήσουν εκεί που γεννήθηκαν. Οι μετανάστες που έγιναν αποδεκτοί σε περιοχές που αποκαλούν τώρα και χώρες που αποκαλούν πατήδες τους, αλλά σε πολλά μέρη αυτό δεν ισχύει ακόμα. Ε, είναι αλήθεια ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθούν να παραβιάζονται σε όλο τον κόσμο και εδώ στην Ευρώπη ακόμα. Και σε κάποιες χώρες η κατάσταση επιδεινούται. Όμως τα καλά μαντάτα είναι ότι τίποτα ε, δεν είναι αναπόφευκτο. Μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στη θετική αλλαγή και όλοι έχουμε συμφέρον να το κάνουμε αυτό. Κάθε άτομο, κάθε χώρα, κάθε θεσμός έχει επιλογή σαφή να κάνει και εγώ πιστεύω στην δύναμη, τη διάδοση των θετικών αποτελεσμάτων που μπορούν να διαδοθούν. Και όταν διηγούμεθα καλέ ιστορίε μπορούν να δώσουν κίνητρα. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάνει επιλογή. Αυτό το κοινοβούλιο γιόρτασε και υποστήριξε Ανθρώπου όπω τον Ντένι Μακουέμπε και την Τάνια Μουράτ. Του τίμησε ε, επί σειρά ετών και κατά τη διάρκεια των στιγμών που είχαν ανάγκη. Με το πρόγραμμά μα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερασπιστήκαμε ανθρώπου σαν και εσά όταν δικαζόσασταν, όταν η ζωή σα και η οικογένειά σα απειλήθηκε. Μαζί συνεργαστήκαμε και δημοσία και σιωπηλά, κατηδίαν κάποιε φορέ, να πετύχουμε απελευθέρωση ακτιβιστών τη κοινωνία των πολιτών και ηγετών τη αντιπολίτευση. Το κάναμε μερικού μήνε σε μια χώρα όπω είναι το Τζερμπαϊτζάν. Και όπω εξακολουθούμε να κάνουμε κάθε μέρα, παντού, ε, σε όλο τον κόσμο, σε χώρε που είναι κοντά στι δικέ μα χώρε και σε αυτέ που είναι απόμακρε. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την οργάνωση για την Ισλαμική Συνεργασία για πρώτη φορά για να περάσουμε ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το ΙΕ για να δημιουργήσουμε μηχανισμό ε, λογοδοσία, διεθνούς λογοδοσίας για το Μιανμάρ. Ένα παράδειγμα, αλλά όπω είπε και ο Αντώνιο, το έργο μας συνεχίζεται στις πατρίδες μας, οι κοινωνίες μας εδώ στην Ευρώπη δεν είναι τέλειε και υπέχουμε καθήκον και για λόγους αξιοπιστίας Συνεχώ να εστιαζόμεθα επί της καταστάσεω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό της υπήρου μα. Θα ήταν υπέροχο αν τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούσαν να επιτευχθούν και να εφαρμοστούν άπαξ διαπαντό, αλλά δεν πηγαίνουν έτσι τα πράγματα και στη ζωή, στην πραγματικότητα, ποτέ δεν επιτυχάνονται δια ε, οι ε, Πάντα είναι ένα εργοτάξιο τα ανθρώπινα δικαιώματα και κάθε γενιά έχει συγκεκριμένη ευθύνη. Σε δύσκολους καιρούς, χαλεπούς καιρούς όπως τώρα, ε, νομίζω ότι η ευθύνη μας είναι να αποφύγουμε ένα λάθος. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε έναντι της ιδέας ότι αυτή η διακήρυξη ανήκει σε μια άλλη εποχή ή ίσως να ισχύει μόνο για μερικές χώρες, ότι είναι κάτι από το παρελθόν αποκαλείται ε, Οικουμενική Διακήρυξη για ένα λόγο. Διότι εκπρόσωποι από όλα τα μέρη του κόσμου συναντήθηκαν, ενώθηκαν και συμφώνησαν επί αρχών που δεν ανήκαν σε έναν πολιτισμό και σε μια κουλτούρα. Επεράσαμε, είχαμε περάσει από τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ανθρώπινη ιστορία. Και εμεί οι Ευρωπαίοι είχαμε τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή την καταστροφή μετά τον πόλεμο. Και όλο ο κόσμο τότε βρήκε το θάρρο να μαζευτεί, να συναθριστεί, να βρει κάποιο κοινό τόπο μετά από την πιο μεγάλη καταστροφή τη ιστορία. Να βρει κάποιο ε, κοινό τόπο πέρα από ιδεολογικέ, θρησκευτικέ, πολιτισμικέ διαφορέ και να ενωθεί. Σήμερα πρέπει να βρούμε εκ νέου αυτό το πνεύμα τη παγκόσμια ενότητα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει κάτι που μα δένει σαν ανθρώπου, σαν ανθρώπινα όντα, πέρα από τι διαφορέ που έχουμε και τι διαφωνίε μα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτή η οικουμενική διακήρυξη του ΟΗΕ, ε, το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, ΟΗΕ και όλοι οι νόμοι επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει δεν είναι περιορισμός, δεν αποτελούν εμπόδιο κατά της επίτευξης των συγκεκριμένων εθνικών στόχων και συμφερόντων. Όταν μαζευόμαστε, το αντίθετο συμβαίνει. Αυτές οι αρχές, αυτό το κοινό έδαφος είναι το θεμέλιο για τη συνύπαρξή μας και ο μόνος τρόπος που έχουμε ούτως ώστε να διαφυλάξουμε, να προωθήσουμε τα εθνικά συμφέροντα και να αποφύγουμε και να προλάβουμε ακόμα μια καταστροφή. Ε, ε, μετά από 70 χρόνια πρέπει να επιστρέψουμε στο πνεύμα του 1948 και θα πρέπει αυτή την οικουμενική διακήρυξη να την έχουμε στο επίκεντρο των καθημερινών προσπαθειών. Θα κλείσω λέγοντας ότι δεν είναι μια επέτειος, δεν είναι μια ανάμνηση, ένα μνημόσυνο θέλετε, είναι ένα μανιφέστο για σήμερα η οικουμενική αυτή διακήρυξη. Πρέπει να είναι ο φάρος για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι και για τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, κυρίως για την καθημερινή δουλειά που μας βοηθάτε να επιτελούμε. Ευχαριστώ. I am delighted to... Είμαι ιδιαίτερο ευτυχή που μπορώ να μεταφέρω τι ε, καλύτερε ευχέ μου για την, επέτειο, την 70η επέτειο από ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα ε, που είναι η Οικουμενική Δίκαιωση των Οποίων Δικαιωμάτων. Ένα κείμενο ορόσημο που διακηρύσει το κοινό μα όραμα για την ανθρώπινη πρόοδο και ευημερία. Όμω, παρά τα ωφέλη που είχαμε το 1948, εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπάρκειε. Βλέπουμε επικίνδυνη διάβρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των δημοκρατικών αρχών του κράτου δικαίου πρόσφυγε, μετανάστε, μειονότητε, όλο και περισσότερο το μίσο και επιθέσει εναντίον του. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δέσμευσή μα ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ε, συνανθρώπων μα. Είναι ένα σκοπό. σημαντικό για την προώθηση τη ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη για την σταθερή εταιρική σχέση που έχουν συμπήξει αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνω την Προεδρία στον κύριο Παντζέρη. Τον ευχαριστώ για τη μεγάλη συνεισφορά του, την προσπάθεια που κατέβαλε για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, τον κύριο Ταγιάννη Ευχαριστούμε και το Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κουτιάζη το μήνυμα που μας έστειλε και την είπα την εκπρόσωπο την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη που άνοιξαν τις εργασίες αυτής της συναντήσεως με σημαντικά λόγια. Θα ήθελα να ποτίσω φόρο τιμής στην προσπάθεια που καταβάλουν για να δίνουν προτεραιότητα στο αιματολόγιο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και το ΙΕ την προστασία και προώθηση των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαίρομαι που ανοίγω το πρώτο πάνελ της διασκέψεως υψηλού επίπεδου με φιλοξενούμενους επιφανείς αξιοσημείωτους για τις προσπάθειες που κάνουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όπως ήδη υπόθηκε, η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενέπνευσε πάνω από 80 διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και συντάγματα πολλών χωρών κάνουν ρητή μνήα, ρητή αναφορά στη διακήρυξη αυτή την οικουμενική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται περί ενό εγγράφου που έχει μεταφραστεί περισσότερο Μεταφράσεις πάνω από 55 μεταφράσεις έχουν γίνει σε διάφορες γλώσσες. Τι τελευταίε δεκαετίες έγινε πολλή δουλειά για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από διάφορα κινήματα, από διάφορε κυβερνήσει και από την κοινωνία των πολιτών. Αυτή η συλλογική δράση ήταν απαραίτητη για την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να πω ότι παρά τις σημαντικές προόδους για τη μείωση της φτώχειας της δεκαετίας του 90 οι ανισότητες εντός των χωρών έχει αυξηθεί και εκεί όπου η ανισότητα μειώθηκε επιτυχώς παραμένει σε ένα επίπεδο σημαντικό υψηλό. Το πρόβλημα της ανισότητας απειλεί να αποδυναμώσει την πρόθεση και τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Οικουμενικής Διακήρυξης. Γι' αυτό πιστεύω ότι η μείωση των ανισοτήτων και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έπρεπε να πηγαίνουν χέρι με χέρι και να είναι ενιαία η μάχη που δίδεται γι' αυτά. Και αυτό μεταξύ άλλων είναι στους βασικούς στόχους του θεματολογίου της Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εργάστηκαν συνεργαζόμενα για να προωθήσουν έναν κόσμο που θα εδράζεται επί κανόνων, επί διεθνούς δικαίου και επί πολυμερούς συνεργασία και προσεγγίσεως. Και δική μα ευθύνη περισσότερο ποτέ είναι καθημερινά να ε, το πυρήνα των διεθνών συνθήκων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι νομικά δεσμευτικά αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα νέες προκλήσεις. Σήμερα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και στρατηγικές ε, προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Θα θέλαμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα καθολικά, είναι κρίσιμη σημασία σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Γιατί είναι σημαντικό να προστατεύσουμε και να, προωθήσουμε, να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε του προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποια είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γιατί είναι σημαντική. Ε, Πώ να προστατεύσουμε καλύτερα όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένη και τη πρόκληση τη ανισότητα. Πώ να προσπιστούμε και να προωθήσουμε τον καλύτερο τρόπο μια τάξη που βασίζεται επί κανόνων με πολυμερή προσέγγιση στο τέλο, με πλουραλισμό. Να ενισχύσουμε τη διεθνή ευθύνη και την καταπολέμηση κατά τη ατιμορρησία. Γι' αυτό είναι σημαντικό στον κόσμο. Και τέλος, είναι σημαντικό να προωθήσουμε αφηγήματα θετικά στον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικά. Εύχομαι σε όλου μια καρποφόρα συζήτηση. Όπως υπόθηκε, έχουμε σημαντικούς φιλοξενούμενους που θα σα παρουσιάσω σιγά σιγά. Δίνω το λόγο. Δέκα λεπτά ο καθένας θα έχει. Στο Μισελ Μπασελέ είπατε εκπρόσωπο το ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Uh, thank you, Την κυρία Μπασελέ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πιέρα Αντώνιο Παντσέρη, πρόεδρε τη Υποεπιτροπή Ανθρωπιδευμάτων Κοινοβουλίου, κύριε Ευρωβουλευτέ, κύριοι Εθνικοί Βουλευτέ από 28 Εθνικά Κοινοβούλια, εξοχότατε, ε, ε, κύρια ε, Αντιπρόεδρε τη Επιτροπή και είπατε επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι παρούσα μεταξύ ενό διακεκρωμένου και σεβαστού πάνελ. Και το θέμα μου είναι πώ μπορούμε να προωθήσουμε ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη και στον κόσμο για να υποστηρίξουμε την, οικονο, την οικουμενική διακήρυξη. Ερνάν Σάντα Κρούθ, ε, που είναι από τη χώρα μου και από τους συντάκτες, έλεγε ότι η έγκριση ε, της οικουμενικής διακήρυξης είναι ένα πραγματικά ιστορικό γεγονός ε, όπου και επιτεύχθηκε συνένεση σε ό,τι αφορά το ότι ο άνθρωπος έχει ύπατη, υπέρτατη αξία και η αξία δεν καθορίζεται από μία εξουσία. Μόνο και μόνο από την ύπαρξή του καθορίζεται αυτή η αξία και επομένως έχει το αναπαλωτρίο το δικαίωμα του να ζει ελεύθερος από καταπίεση, να μπορεί να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Αυτά είχε πει ο Ερνάν και η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οδήγησε σε τεράστια βήματα πρώτη την ανθρωπότητα τα τελευταία 70 χρόνια στον τομέα της υγείας, εκπαίδευσης, της ειρήνης, της βιώσιμης ανάπτυξης είχε οδηγήσει και σε μικρότερη περιοθεροποίηση των ε, μειονοτήτων, επανεπιβεβαίωση του δικαιώματο στην ισότητα, ε, κατά τη τυραννία, κατά τη εκμετάλλευση, ε, πρόσβαση σε βασικέ υπηρεσίε, οικονομικέ δυνατότητε και ευκαιρίε. Πρέπει κανεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη των επιτευγμάτων σε μια εποχή που πριν από δεκαετίε ήταν το επίκεντρο οικονομική καταπίεση και φρίκη του ολοκαυτώματο. Ε, η δικαιοσύνη προωθήθηκε και έχουμε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο ε, με επίκεντρο το κράτος δικαίου, σταθεροί θεσμοί, ε, ελεύθερα μέσα ενημέρωση, ανοιχτή κοινωνία, ένας χώρος ανάπτυξης των ιδεών, κοινωνίες πιο αλληλέγγυες, υπάρχει μεγαλύτερη ένταξη, μεγαλύτερο σεβασμός, οι δράστες των διαφόρων εξώπνων πράξεων διώκονται. Υπάρχει δυνατότητα καλύτερης επανόρθωσης πλέον ε, και η λογοδοσία έχει βελτιωθεί. Ενισχύονται τα δικαιώματα και λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ε, των ανθρώπων. Όταν θα μπορούσε κατά το παρελθόν ε, να υπάρχει αυτή η τυραννία, την έζησαν οι παππούδες μας, τώρα βλέπουμε μια αλλαγή μετά την Οικουμενική Δικαίωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πολλές διατάξεις τις έχουν δε ε, συμπεριληφθεί και στο νόμο αλλά είναι και πράξη. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο δεσμευτικών συνθήκων ε, από τους διεθνείς δικυβερνητικού οργανισμούς. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι στηρίζουν ε, τις δεσμεύσεις που κάνουν τα διάφορα κράτη. Όταν καθημερινά εργάζομαι και βλέπω τις σειράξεις που υπάρχουν ακόμη, δύσκολο είναι κανείς ε, να ε, εστιάσει μόνο στα θετικά αυτής της 70 όμως υπάρχουν πολλά θετικά. Πρόοδος έχει επιτελεστεί, αλλά πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν. Αγαπητοί λοιπόν φίλοι, οι αξία των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό. Συνεχίζουν ε, να προωθούν τεράστιες αλλαγές. Όλοι όμως αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε ένα ταραγμένο, πολλωμένο κόσμο σήμερα που γιορτάζουμε την 70η επέτειο της οικονομικής διακήρυξης ε, υπονομεύεται η ειρήνη πρόοδος ε, προς κοινού στόχους ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν σειράξεις, αντιπαραθέσεις που δημιουργούν μεγάλη οδύνη, εκτοπίζουν πληθυσμούς η ισότητα ανδρών και γυναικών, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΟ και τα δικαιώματα εθνικών ή ε, θρησκευτικών μειονοτήτων. Τίθεται υπό αμφισβήτηση, συρρυκνούνται ο κοινωνικό ιστό και πολλοί υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων διώκονται, ε, απειλείται η ζωή του, ε, θανατώνονται. Επίσης, τα σεξουαλικά αναπαραγωγικά δικαιώματα δεν είναι παντού αναγνωρισμένα και βλέπουμε οπισθοδρόμοι σε σχέση με την πρόοδο των προηγούμενων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχουν ε, ε, τα θεμέλια ε, για την προσέγγιση των δικαιωμάτων, η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία της έκφρασης. Βλέπουμε ότι διαβρώνονται αυτά σε μερικές χώρες. Υπάρχει ρητορική μίσους κατά μεταναστών, κατά μειονοτήτων Επομένως, είναι σημαντικό να συνεχίσει η πρόοδος ε, παντού ε, σε ό,τι αφορά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην έχουμε οπισθοδρόμηση ώστε όλες οι κοινότητες να συμπεριφθούν. Η Ρωμά, για παράδειγμα, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι άποροι, σε μια κοινωνία που τα δικαιώματά τους ε, θα είναι σεβαστά. Υπάρχουν στον πλανήτη μας ανισότητες που απειλούν το στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης ε, να τους ε, ε, κάνουν να φαίνονται μακρινοί. Έχουμε την αλλαγή του κλίματος που εντείνεται και δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από κοινού λοιπόν έχει έρθει να αντιμετωπίσουμε την ώρα της αλήθειας και έχουμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τη σημασία της πολυμερούς διακυβερνητικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της δίνης που προκαλούν όλες αυτές οι διεθνείς προκλήσεις. Πρέπει να εφαρμόσουμε από αποφάσεις ε, διεπόμενη από τη σαφήνεια ε, του νόμου, τη νομοθεσία για το ανθρώπινο δικαίωμα. Όταν μιλάμε για εθνικισμούς, αλλαγή του κλίματο, μετανάστευση, οικονομικέ και κοινωνικές ανισότητες, ε, δικαστική ανεξαρτησία, ελευθερία έκφραση, μαζικές παρακολουθήσει, τεκτή νομοσύνη κτλ. Η ζωτική σημασία είναι να έχουμε τα το, ως το μεγαλύτερο ζωτικό χώρο για δημόσια έκφραση και συμμετοχή και στο επίκεντρο βέβαια είναι τα αστικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά δικαιώματα. Πρέπει ε, όλοι μας να συνεργαστούμε προς αυτό το στόχο στο πλαίσιο ε, των διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου ή των δικαίου δικαιωμάτων. Μεγάλες οι επιτυχίες ε, μέχρι στιγμής και ευεργετικές για όλους. Όμως υπάρχουν έντονες πιέσεις σήμερα και πρέπει να συνεχίσουμε να σεβόμαστε αυτή την νομοθεσία. Μέρο της πρόκλησης είναι οι διεθνεί αυτοί κανόνες, διεθνή πρότυπα να γίνουν πιο κατανοητά αποδεκτά από τους χαράκτες πολιτικής ε, μεταδίδοντας ακριβώ ε, τους ε, τρόπους με τους οποίους θα μπορεί να ωφεληθεί ο κάθε άνθρωπος. Είπε και η Φεντερίκα Μογκερίνη Έχουμε και το Σταύρο Λαμπρινίδη μαζί μας ε, και σίγουρα πρέπει να καταγγέλουμε τα απαράδεκτα αλλά πρέπει να δείχνουμε και τα καλά, ε, να προωθούμε τα θετικά ε, που μπορούν να προκύψουν. Ισχυρές κοινωνίες, πιο βιώσιμη ανάπτυξη, πιο τελεσματική πρόληψη συγκρούσεων. Θέλουμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός όλοι μας, κυβερνήσεις, κοινοβούλια, κοινωνία των πολιτών, ε, το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ιδιωτικό τομέας, άνδρες, γυναίκες και παιδιά πρέπει ε, να καταπολεμήσουμε ε, τη δαιμονοποίηση ε, των μεταναστών, των μειονοτήτων και άλλων ε, ομάδων. Πρέπει τη ρητορική μίσους να την απορρίψουμε. Στρεφόμενοι πάλι στην οικονομική δικαιοσύνη των δικαιωμάτων, η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια, αυτό είναι το έρισμα στρέφομαι και βλέπω μια Ευρώπη που έχει το στένος, έχει το κουράγιο να συνεχίσει να δημιουργεί περισσότερα επιτεύγματα, διατηρεί, αναβαθμίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική πρόοδος, ε, η αλληλεγγύη είναι μεγάλες ε, δυνάμεις. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτά που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές στο ψηφιακό κόσμο και να διέπουν επίσης όλες τις δημόσιες πολιτικές. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαλόγου, να ενισχύσουμε την κουλτούρα του αλληλοσεβασμού να ενστερνιστούμε τη διαφορετικότητα. Σήμερα έχουμε και την ημέρα για τη δουλειά των παιδιών. Ας τους δώσουμε λοιπόν ε, μια σημαντική κληρονομιά, ώστε τα παιδιά στην περιοχή αυτή, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη, ε, και τα παιδιά αυτών να μεγαλώσουν ε, έχοντας πλήρη πίστη στην ακαιρεότητα, στο αναπαλωτρία το δικαίωμα όλων των ανθρώπων όπως αυτά αναγνωρίστηκαν πριν από 70 χρόνια. Είναι η ελευθερία, η ειρήνη και η δικαιοσύνη στον κόσμο αυτά τα θεμέλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πραγματικά για τη σημαντική αυτή συνεισφορά. Να δώσω το λόγο στην Τάμφα Μπενσούντα από το Εθνές Ποινικό Δικαστήριο, συντονίστρια. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Your Excellencies, fellow ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου εκ των προτέρων να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κύριο Ταγιάννη, όπως και τον Πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Παντζέρη, για την οργάνωση αυτής της συνάντησης και για την πρόσκλησή τους. Είναι τιμή μου που μπορώ να απευθυνθώ σε εσά σε αυτό το ε, εντυπωσιακό χώρο και μάλιστα μαζί με τόσους σημαντικούς ομιλητές που συλλογικά δείχνουν την τεράστια προσπάθεια γίνεται για την διεθνή ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σημερινή εκδήλωση φυσικά αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένα χρονικά σημεία όπως τα 100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 70 χρόνια από την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως επίσης και τα 20 χρόνια από την δημιουργία του συνθήκης της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλα αυτά δείχνουν την βελτίωση των διεθνών επιπέδων προστασίας και προάσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι ένα δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μια στενή ερμηνεία. Η σημασία του όμως για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Ε, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανθρωπότητα προσπαθούσε να σηκωθεί μετά από την αφάνταστη καταστροφή και δυστυχία και την τεράστια βία που είχε υποστεί. Υπήρξε μια προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους δράματα ένωσαν τα χέρια τους για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο κόσμο, να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να θέσουν ένα τέλος στην ατιμορρησία. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι πρώτες διεθνείς συμφωνίες για το ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές ποινικό. 70 χρόνια μετά η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει το συνταγματικό θεμέλιο της αναγνωρισμένης πλέον αυτής προσπάθειας. Ε, μετά από τις ε, δίκες των εγκληματιών στην Ιρεμβέργη και στο Τόκιο δημιουργήθηκε ένα παράδειγμα για να, μην, για να ελέγχονται πλέον αυτοί οι οποίοι διαπράττουν τέτοιου είδους φρικτές πράξεις. Οφεληθήκαμε φυσικά επίσης ε, και από μια αίσθηση ανάγκης μετά τον ε, ψυχρό πόλεμο και μετά από την ε, γενοκτονία στη Ρουάντα όπως και στην πρώην Ιουκοσλαβία είδαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη αν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τον μη σεβασμό της δεν τιμωρηθούν. Το Διεθνές Ποινικό δημιουργήθηκε λοιπόν μετά από τη διάσκεψη της Ρώμης το 1998 ε, σαν ένα είδος ε, συνειδητοποίησης ε, και συγκεκριμένοποίηση της τεράστιας προσπάθειας, της συλλογική προσπάθειας για να τεθεί τέλος στην ατιμορρησία των ενόχων από την διεθνή κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε και πολιτικά και πρακτικά πολύ σημαντικό ρόλο για να γίνει το διεθνές ποινικό λειτουργικό. Ε, το δικαστήριο επίσης υποστηρίζεται και από τις 27 χώρες μέλη που είναι φυσικά χώρες που συμμετέχουν και στην Σύμβαση της Ρώμης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μαζί με ένα ανεξάρτητο λοιπόν και μόνιμο διεθνές ποινικό δικαστήριο η συνθήκη της Ρώμης στην ουσία δημιουργεί ένα αλληλένδετο σύστημα ε, διεθνούς ποινικού δικαίου το οποίο εδράζεται ε, στις βασικές αρχές της συμπληρωματικότητας και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο φυσικά διμερές και σε επίπεδο πολυμερές το διεθνές ποινικό το οποίο είναι ο πυρήνας θα έλεγα αυτής της προσπάθειας με τη δική μου υπηρεσία ως κινητήρια δύναμη προσπαθεί να διώξει αυτούς οι οποίοι παραμένουν ατιμόρυτοι για φρικτά εγκλήματα τα οποία δυστυχώς ακούμε καθημερινά στον κόσμο. Ε, στον σημερινό κόσμο βλέπουμε την φρίκη να μολύνει και γειτονικέ χώρες και να περνάει και από τη μία ήπειρο στην άλλη και να οδηγεί στην καταστροφή εθνικών θησαυρών και πόλεων. Κάθε ε, ε, μέρα, κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά, γυναίκες και άνδρες είτε επηρεάζονται απλά αρνητικά είτε πέφτουν θύματα αυτής της απαράδεκτης βίας όπως και της σωματεμπορίας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν η υπηρεσία μου προσπαθεί να αποδώσει όλο και περισσότερο και εξετάζουμε ε, τέτοιου είδους πιθανά εγκλήματα σε όλες τις περιοχές του κόσμου, από την Ουκρανία, την Ιγυρία, την Κολομβία, τη Βενεζουέλα, στην Παλαιστίνη, τις Φιλιππίνες και τη Μιαμάρ, Μπαγκλαντές. Ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αν οι καταστάσεις αυτές δικαιολογούν και τεκμηριώνουν το να ξεκινήσει μια δικαστική διαδικασία και προσπαθώντας ε, να πιέσουμε τις εθνικές δικαστικές αρχές να διώξουν τα εγκλήματα αυτά. Και ε, επίσης έχουμε ζητήσει έτσι, να ώστε να μπορέσουν οι δικαστές του Διεθνούς Ποινικού να δραστηριοποιηθούν και στο Αφγανιστάν. Έχουμε ε, δραστηριοποιηθεί και στη Γεωργία και στο Μπουρούντι και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και έχουμε δώσει εισαγγελικές παραγγελίες και για την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία και τη Λιβύη και την Ουγκάντα όπως και την ακτή του Ελεφαντόδοντος. Ταυτόχρονα ε, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε διώξεις και στην Δημοκρατία του Κονγκό όπως και στο Μαλί και έχουμε επίσης εκδώσει και εντάλματα σύλληψης για 15 ε, προσώπα τα οποία θεωρούμε ότι ε, βάσιμα μπορεί να κατηγορηθούν για εγκλήματα τα οποία καλύπτονται από τη συνθήκη της Ρώμης. Νομίζω ότι από τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε και σε επίπεδο τεκμηρίωσης και σε επίπεδο διώξεων είναι χρήσιμες για τη διεθνή δικαιοσύνη. Παραδόθηκε στην δικαιοσύνη και στο Διεθνές Ποινικό ο κύριος Γέκατομ, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Βέβαια ε, η επιδίωξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Ε, το βάρος της παρέμβασής μας εξαρτάται από το επίπεδο πολιτικής, διπλωματικής, λειτουργικής και οικονομικής στήριξης την οποία λαμβάνει από τα κράτη-μέλη και όλους τους άλλους εταίρους. Απαιτείται η συνεργασία έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε πλήρως την ύπαρξη του διεθνούς ποινικού και άλλων διεθνών μηχανισμών δικαιοσύνης. Η συνεργασία απαιτείται για να αυξηθεί ο αριθμός των κρατών που συμμετέχουν στο διεθνές ποινικό. Η συνεργασία απαιτείται επίσης για να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες στις διάφορες χώρες να αντιμετωπίζουν τα φρικτά εγκλήματα σε εσωτερικό επίπεδο και να κλείνουν το λεγόμενο ρήγμα της ατιμορρησίας μέσω της συλλογής εμπειρογνωμοσύνης και ανταλλαγής πληροφοριών. Η διεθνή ποινική δικαιοσύνη είναι μια παγκόσμια προσπάθεια που θα ωφελήσει το σύνολό της ανθρωπότητας. Όλοι έχουμε την ευθύνη να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε τους στόχους αυτούς όπως και οι διεθνές ποινικέ δραστηριότητες, εγκληματικές δραστηριότητες μάλλον, προσαρμόζονται στον ψηφιακό και παγκοσμιωμένο κόσμο, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Προσπαθούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να χρησιμοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων καιρών, την ικανότητά μας να παρουσιάζουμε, να συλλέγουμε και να παρουσιάζουμε ε, αποδείξεις που να βασίζονται στις σύγχρονες τεχνολογίες. Σαν παράδειγμα σχετικά με την έκδοση εντάλματος για τον Μαχμούντ Μουστάφα Αβερφάλι. εμείς χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ και βίντεο και τα κοινωνικά μέσα, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά κοινωνικά μέσα. Μπορούμε να κάνουμε όμως πολύ περισσότερα. Πολλές οργανώσεις έχουν αρκετές γνώσεις και προσπαθούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Εκεί όπου εμείς δεν μπορούμε να δράσουμε ε, τότε τα δεδομένα και τα ψηφιακά στοιχεία που συλλέγονται από άλλες οργανώσεις μπορεί να είναι κρίσιμα για την επιτυχία μας. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη συνεργασία μας με, τους, ε, με τις οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές μετά από ένα σύμβαν. Αυτές οι βελτιωμένες μορφές συνεργασίας και οι... Ε, κατανομή, μάλλον η, η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να μας βοηθήσει να συλλέξουμε τις ζωτικές αποδείξεις και να περιορίσουμε τον χρόνο που απαιτείται. Και τέλος είμαστε υποχρεωμένοι σε διεθνές επίπεδο να πάρουμε βήμα, να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να είναι υπόλογοι τελικά όλοι όσοι παραβιάζουν ε, την διεθνή ποινική, τις ε, ρυθμίσεις. 70 χρόνια μετά λοιπόν από τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, μετά από αρκετά χρόνια μετά τη δημιουργία του διεθνούς ποινικού θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι ε, όλοι μπορούμε να παραδεχθούμε ότι ε, οι άνθρωποι έχουν τα δικαιώματα αυτά όλοι χωρίς καμία εξαίρεση και πρέπει να τα προστατεύσουμε τα δικαιώματα αυτά. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τα θύματα των χειρότερων παραβιάσεων να υποφέρουν σιωπηλά. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτοί οι οποίοι διαπράττουν αυτά τα φρικτά εγκλήματα να διαφεύγουν της τιμωρίας. Όπως και η κυρία Μογκερίνη μόλις μας είπε, ή μάλλον μας είχε πει στις 13 Σεπτεμβρίου ε, νωρίτερα είναι ένα πράγμα να νιώθει κανείς ε, ε, ανήμπορος και αδύναμος αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιδιώξουμε να τιμωρηθούν αυτοί που προκάλεσαν αυτή την κατάσταση και είναι απαραίτητο αυτό για να θεμελιωθεί εκ νέου η ειρήνη στον κόσμο και πράγματι θα πρέπει οι διεθνείς αυτές οργανώσεις να γίνουν ισχυρότερες και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πολυμερές ακόμα πιο ισχυρό από το σημερινό. Έτσι θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε το σύνολο της ανθρωπότητας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αντιμετωπίζεται σαν ένα μέσο προσφυγής για το σύνολο της ανθρωπότητας. Ε, στο προήμιό μας, στο προήμιο του κανονισμού λειτουργία μας λέγεται ότι όλοι οι λαοί του κόσμου έχουν κοινά μεταξύ τους και αυτό το ευαίσθητο μοσαϊκό μπορεί να διαρριχθεί μέσω της διάπραξης σημαντικών εγκλημάτων. Εμείς λοιπόν ευχαριστούμε και εκτιμούμε την υποστήριξη την οποία παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως επίσης και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πιστεύουν στο διεθνές ποινικό και θεωρούν ότι είναι ένα καλό μέσο για την προστασία του προσώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όσο όμως συνεχίζουμε εμείς ενωμένοι να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα της ατιμορρησίας είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να περάσουμε σε έναν κόσμο με λιγότερες σειράξεις έναν κόσμο με περισσότερο σεβασμό για τους κατοίκους της γης αυτής σε όλες τις γωνιές αυτού του πλανήτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να συνεχίσουμε την συνεργασία με όλους σας. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Σταύρο Λαμπρινίδη, ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Uh, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε Αντώνιο. Αγαπητοί φίλοι, είμαστε ανθρώπινα όντα, δεν είμαστε ζώα. Δεν μπορείτε να με κλωτσίσετε. Δεν μπορείτε να το σκοτώσετε, δεν μπορείτε να με φυλακίσετε. Δεν μπορείτε να με αντιμετωπίσετε σαν ζώο επειδή ε, δεν σας αρέσω. Και αυτό γιατί έχω ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το πιο απλό πράγμα που ανέφερε εδώ και 70 χρόνια η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει αυτή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οποιοδήποτε πολιτισμό και αν δείτε, οποιαδήποτε θρησκεία, οποιοδήποτε σύστημα ή περιοχή στον κόσμο θα δείτε ότι αποτελεί τον πυρήνα του συστήματο στο οποίο πιστεύουν. Δεν υπάρχει κανένα μέρο στον κόσμο που η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ιστορικά δεν αποτελεί ένα τμήμα τη φιλοσοφία του περιζωή. Παρ' όλα αυτά, αυτοί που θέλουν να παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αυταρχικοί στον κόσμο, ποτέ δεν του άρεσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στου δικτάτορε δεν του άρεσαν τα δικαιώματα. Αλλά εκείνοι που θέλουν να κάμψουν τη βούληση του λαού τους, να, κα, να κάμψουν τη βούληση των θεσμών και να τα καθυποτάξουν και τις περιφέρειες και τις περιοχές να τις καθυποτάξουν, δεν αντέχουν την ανοχή, δεν αντέχουν τη συμπερίληψη, δεν αντέχουν το κράτος δικαίου. Προσπαθούν να μας διχάσουν, να μας κάνουν να μισήσουμε εμέν τους δε, προσπαθούν να μας κάνουν να βλέπουμε ένα τον άλλον με μάτια μίσους με το μίσος ζώων. Θα τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Θα τους αφήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι. Και εμείς επί σειρά τον λέμε όχι. Και λέμε νο, ε, όχι συγγνώμη παρά τις ατέλειες μας. Και λέμε όχι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο προθώντας τα δικαιώματα. Λέμε όχι παρά το γεγονός ότι εκείνοι που ιδεολογικά είναι ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικά ε, στρέφονται κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι καλοί στην εξαγωγή κακών αφηγημάτων και κακών πρακτικών προς τους άλλους. Πολύ συχνά έχω ακούσει τις επισκέψεις μου να μου λένε γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτεται το θέμα των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων και των λεσβιών. Κοιτάξτε τις δημοσκοπήσεις στη χώρα μας. Δεν αρέσουν στον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί μιλάτε για θανατική ποινή. Κοιτάξτε τι λέει η κοινή γνώμη στις δημοσκοπήσεις στη χώρα μου. 90% του κόσμου την υποστηρίζει θανατική ποινή. Γιατί ε, θίγεται αυτά τα δυσάστα θέματα. Γιατί να μιλήσουμε για παραδάκι, για χρήμα, αυτά που μας ενώνουν. Η απάντησή μου σε αυτό πολύ συχνά ποια είναι. Αν θέλετε να μιλήσετε μόνο για χρήματα σε λάθο μέρο με λάθο ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι ε, άλλοι που θα τα γνωρίσουν αυτά. Αλλά εμεί έχουμε βγει από τον πιο αιματηρό πόλεμο στον κόσμο, από τι μεγαλύτερες παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 70 χρόνια, αυτή την επέτειο είμαστε η πιο ειρηνική περιοχή στον κόσμο, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, γιατί αποφασίσαμε ότι δεν θα οικοδομήσουμε οτιδήποτε εκτός αν τα θεμέλια είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οτιδήποτε άλλο σε κινούμενη άμμο ε, χτίζεται. Μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή. Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας. Θα πρέπει να συνεργαστείτε και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και υπάρχει και άλλος λόγος. Ποιος είναι αυτός. Ότι ουσιαστικά εκείνος που, όπως είπε Μισελ, για όλους εκείνους τον κόσμο, που είναι απομονωμένοι, καταπιεσμένοι, τους φέρονται σαν ζώα και η κοινωνία των πολιτών, για όλους αυτούς που δίνουν αυτή τη μάχη στον κόσμο, δεν προστατεύει ο καθένας από αυτούς κάποια μειονότητα εδώ και εκεί. Όλοι προστατεύουμε τη δημιουργία ειρηνικών, τεραστίων κοινωνικών συνόλων ειρηνικών, προστατευμένων, διότι κάθε κοινωνία στον κόσμο οικοδομείται βάσει του σεβασμού εκατοντάδων μειονοτήτων. Σε μια αίθουσα που είσαστε η πλειοψηφία λόγω του φίλου σας Φερρυπίν και θεωρείτε ότι εξ αυτού μπορείτε να καταστήλετε, να καταπιέσετε το άλλο φίλο που είναι στην μειοψηφία, είναι στη μειονότητα, στην ίδια αίθουσα, στην πλειοψηφία που κατέχετε Εσεί ο ίδιος, η ίδια μπορεί να είστε μειοψηφία, μειονότητα, λόγω πολιτικών απόψεων, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, λόγω για αντιμετωπίσετε κάποιον άλλο σα ζώο είναι ή λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Τη στιγμή που έχετε την εξουσία της πλειοψηφια και αποφασίζετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εξουσία για να αντιμετωπίσετε κάποιον άλλο σα ζώο, είναι η στιγμή ε, που ανοίγετε την πόρτα της κόλασης την πόρτα για να αντιμετωπιστείτε εσείς σαν ζώο. Διότι όλοι είμαστε μειονότητες και μειοψηφίες. Η Φεντερίκα Μογκερίνη το ανέφερε ότι την 70η επέτειο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με 13 χώρες σε όλο τον κόσμο στη Νέα Υόρκη αποφασίσαμε να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα. Ξέρετε γιατί. Διότι όλοι εκείνοι προσπαθούν να παραβιάσουν τα δικαιώματα επί σειρά ετών μας λένε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απελ, άπελπης προσπάθεια. Όλοι τα παραβιάζουν δικαιώματα και αλλιώς. Γιατί ανακατεύεστε στις υποθέσεις μου. Κοιτάξτε τι κάνετε εσείς Ευρωπαίοι, έχετε και εσείς προβλήματα. Κοιτάξτε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν το λένε αυτό για να πούνε πόσον έχουμε όλοι προβλήματα, προσπαθήσουμε συνεργαζόμενοι να τα λύσουμε. Λένε για να μας πούν αφήστε μας ήσυχου, εσείς, να σας αφήσουμε εμεί ήσυχου πέρα το ότι θέλουν να μας κάνουν να διχαστούμε και να μισούμε μεν τους άλλους, θέλουν να αισθανθούμε απελπισμένοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σαν είναι κάτι που λειτουργεί. Μαντέψτε, λειτουργεί κάθε μέρα. Η Μισελ ε, Μπασαλέ, Φατού Μπενζουμά, κάθε άνθρωπος στην αίθουσα σας το είπε ότι είχαν εμπειρίες, είχαν παραδείγματα που άλλαξε ο κόσμος λόγω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι 13 χώρες το έκαναν αυτό στην αίθουσα στη Νέα Υόρκη. Παρουσίασαν ιστορίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένες ιστορίες. Μέσα από τις ιστορίες είδαμε ότι πρόθεσαν οικονομική ανάπτυξη στη χώρα τους, βιώσιμη ασφάλεια, ή ειρηνικέ κοινωνίε και ε, δικαιώματα γυναικών. Η Τινησία μίλησε συγκεκριμένα για τη νέα τη νομοθεσία κατά τη βία κατά των γυναικών. Πολύ, ε, η πολύ ισχυρή κοινωνία των πολιτών με την κυβέρνηση το επέφερε αυτό. Η Μπουρκίνα Φάσο ε, μίλησε για ένα πρόγραμμα όπου 19 οργανώσεις τη κοινωνία των πολιτών παρακολουθούν το πώς εφαρμόζει ο πρόεδρο την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα για να είναι ισότιμη αντιμετώπιση άνευ διαφοράς. Καταμέτρηση της απόδοσης των επιδόσεων του Προέδρου, με άλλα λόγια. Μέσα από ένα μνημόνιο με πολυσέλιδο εφαρμόζεται αυτό. Συμφώνησε να το προσυπογράψει η κυβέρνηση. Συμφώνησε να ελέγχεται, διότι αποφάσισε η κυβέρνηση ότι δεν φοβάται να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών. Αλλά συνεργαζόμενη την κοινωνία των πολιτών ήταν ο καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη σε αυτή την αίθουσα στη Νέα Υόρκη αναλάβουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Έθνη και με τους ειδικού ηγητές του ΟΗΕ ε, και να έχουμε τις δικές μας πρακτικές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να υποπτεύονται και να ελέγχονται. Ε, δεσμευτήκαμε την εφαρμογή του πολυμερού συστήματος για το κράτος δικαίου όχι, κράτο, όχι ε, κυβέρνηση μέσω νόμου, όχι για εκείνους που θεσπίζουν οποιοδήποτε νόμο ωφελεί αυτούς, ακόμα και αν παραβιάζει η διεθνή νομοθεσία και την καθολική διακήρυξη αυτή. Το κράτος δικαίου που στηρίζουμε. Σε αυτή την αίθουσα δεσμευτήκαμε να συνεργαστούμε την κοινωνία των πολιτών καθημερινά, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Και οι κυβερνήσει διαφωνούν, σα διαβεβαιώ. Ξέρω ότι πολλέ φορέ οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών μου ζητούν να του δω, να συναντηθούν μαζί μου. Δεν είναι για να μου πουν ότι κάνω καλή δουλειά. Συνήθω έρχονται να μου πούν ότι κάτι δεν κάνω σωστά. Και εντάξει, Μπορεί να διαφωνώ. Αλλά ε, η ελευθερία και το άνοιγμα που ανοίγουμε για αυτούς τους φορείς είναι κάτι που μας επιτρέπουν να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να βελτιωθούμε. Σε αυτή την αίθουσα δεσμευτήκαμε. Να βελτιώνουμε συνεχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κανείς δεν είναι τέλειος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγαπητοί φίλοι, μία προειδοποίηση. Κοιτάξτε τι προσπαθούν οι κακοί να μας κάνουν να πέσουμε σε δύο παγίδες θέλουν. Η μία είναι θεωρητική παγίδα και η άλλη είναι ε, ψυχολογική. Ποια είναι η διανοητική παγίδα. Θα μας πείσουν ότι επειδή τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σε επαλπιστική κατάσταση και όλοι είναι ατελείς, γι' αυτό συνεπάγεται ότι όλοι είμαστε ατελείς. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πράγματι αληθεύει ότι κανείς δεν είναι τέλειος σε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν διαφορές όμως μεταξύ εκείνων που έχουν δημιουργήσει ανεξάρτητα δικαστήρια, θεσμούς, ανεξάρτητους θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητο ελεύθερο τύπο, ελεύθερα κοινοβούλια, ανεξάρτητα όπω αυτό, που πάντα προσπαθούν να πιέσουν να βελτιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και απ' την άλλη έχουμε τους άλλους που παραβιάζουν ε, χωρίς αχαλήνοντα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τόσο χρόνο, αφιερώνει κόσμο για να επικρίνει δημοσία και κατηδία, να πολεμήσει, να ασχοληθεί με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το πράττουν χώρες, αλλά να συνεργαστεί με όλες εκείνες τις χώρες που πραγματικά θέλουν να συνεργαστούν μαζί μα να δημιουργήσουν δικαστήρια, να δημιουργήσουν ανεξάρτητε εφημερίδε, ανεξάρτητο τύπο, ανεξάρτητου θεσμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δημιουργήσουν μηχανισμού που δίνουν αξία. Παρακαλώ να συνοψίσω λέγοντα τα εξή. Ανέφερα στην αρχή ότι υπάρχουν κάποιοι στους οποίους δεν αρέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθούν να μας διαιρέσουν, να μας διχάσουν, να μας κάνουν να μισήσουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να αντισταθούμε. Υπάρχει κάτι που είπε ο Μαντέλα και εγώ έχω τη δικό μου ρητό του Μαντέλα όπως όλοι οι άλλοι. Τι είπε και θέλω να παραθέσω, τι είπε ο Νέλσον Μαντέλα. Κανείς δεν γεννιέται μισώντας. Αν μπορείς να μάθεις να μισήσεις, μπορείς να μάθεις και μπορούν να σε διδάξουν πώς να αγαπάς. Έχουμε μάθει πώς να μισούμε. Μας δίδαξαν πώς να μισούμε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Αλλά αν όλοι στην αίθουσα, οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, μέλη των κοινοβουλίων, αξιωματούχοι κυβερνήσεων, αυτοί που έχουν το βραβείο Ζαχάροφ, κάτοχοι του βραβείου Ζαχάροφ, αν όλοι φύγουμε έχοντας αναλάβει τη δέσμευση, αυτό να το σταματήσουμε, αυτή τη διολίστηση προς το μίσος, τότε μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο που αγαπάει περισσότερο. Είναι κακή λέξη να το πούμε αυτό. Εστιαστήκαμε σειρά ετών επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα θεωρούμε νομικά μέσα και πραγματικά αληθεύει αυτό. Να τα θεωρούμε σαν νομικά μέσα είναι κάτι που ισχύει. Να λέμε στι χώρε ότι έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν διότι υπέγραψαν δηλώσει και διακηρύξει, αυτό είναι αληθέ. Ισχύει. Ίσως όμως στη διαδικασία κάτι χάσαμε. Μήπως χάσαμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον άνθρωπο, τον απλό άνθρωπο, να τον κάνουμε συντονιστή μαζί μας, να τον συγκινήσουμε, να καταλάβει ο απλός άνθρωπος γιατί αυτές οι αξίες υπάρχουν και είναι πάνω από τους νόμους, είναι, είναι συμπροματικές αξίες του νόμου, δεν θα υπήρχαν οι νόμοι αν δεν υπήρχαν οι αξίες. Εγώ δεν τρέπομαι να μιλώ με πάθο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πω τελικώ από το στόχο είναι να δημιουργήσω περισσότερη αγάπη. Δεν θα επιτρέψω εκείνου που προσπαθούν να μα μισήσουν και να μα διαιρέσουν και να μα διχάσουν να νικήσουν. Δεν πρέπει. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Σταύρο. Η Άμιλι Ράιλι έχει το λόγο διαμεσολαβήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Παντσέρη, αγαπητοί ομιλητές, κυρίες και κύριοι. Με τιμά ιδιαίτερη πρόσκληση να μιλήσω αυτή τη διάσκεψη και θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την προοπτική από την πλευρά του συνηγόρου του πολίτη κατά τους αρτασμούς ε, της απαιτής ε, οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων που έχουμε όλοι, μόνο και μόνο λόγω της ανθρώπινης φύσης μα Αυτό το έγγραφο ποτέ δεν ήταν ο σκοπός του ούτε και ήταν κάτι στατικό. Και συν το χρόνο και όσο αλλάζουν τα πράγματα μπορούμε υπό νέο πρίσμα να διαβάσουμε τα άρθρα του και να δούμε τις νέες ε, πραγματικότητες και προοπτικές. Πάντα έχοντας ε, την πρόκληση ε, του να μην ξεχνάμε τις θεμελιώδεις αξίες. Η δημιουργία του σύγχρονου γραφείου του συνηγόρου του πολίτη στον κόσμο τον τελευταίο αιώνα ήταν ένα από του τρόπου ε, να υλοποιηθούν πολλά από τα δικαιώματα τη διακήρυξη. Γιατί θεμελιώδη ρόλο του διαμεσολαβητή είναι να προστατεύει του πολίτε από κατάχρηση εκ μέρους ε, της ε, κρατικής εξουσίας όταν ε, εφαρμόζει τους νόμους και τους κανονισμούς και δημιουργεί μια ισότητα αμβλύνοντας την ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ πολιτών και κράτους. Έτσι μπορούν με την ήπια δύναμη να εφαρμοστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα με την συμμόρφωση προς τις συστάσεις του διαμεσολαβητή. Έτσι λοιπόν αυτή η ήπια δύναμη κατατρεφτίζεται σε εμά όπως την προέβλεπε η Οικουμενική Διακήρυξη και σίγουρα αν ε, δεν, γίνεται, δεν λαμβάνεται υπόψη το έργο μας αυτό είναι ένα καμπανάκι για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση προς θεμελιώδεις ε, αξίες και δικαιώματα. Διετέλεσα σύμβος του πολύ στην Ιρλανδία και τώρα είμαι Ευρωπαία Δισομελαβητρία. Πολλές φορές δεν επικαλούμε τον όρο ανθρώπινα δικαιώματα όταν παρουσιάζω μια πρόταση στα ε, κρατικές αρχές γιατί πολλές φορές αυτή η ρητορική πολλές φορές γίνεται αντιληπτεί ω κάτι δύσκολο και δαπανηρό από τα κρατημελικό ακόμα λοιπόν, και αν υπάρχουν καλύτερε προθέσει. Καλύτερα λοιπόν να μιλά κανεί για διαδικαστικά κενά ή διοικητικά ασφάλματα, ακόμη και αν το τελικό αποτέλεσμα είναι να ε, πραγματοποιηθεί ε, κάτι πολύ σημαντικό για τον πολίτη, ένα βασικό του δικαίωμα, στέγαση, κοινωνική προστασία, υγειονομική περίθαλψη ή ε, κάποιο άλλο ευεργέτημα δυνάμει τη κοινωνική διακήρυξη. Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα εμπίπτουν στην τα των εθνικών κρατών μελών και όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι καταγγελίε, οποίε εγώ λαμβάνω, είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Πολλέ φορέ αφορούν τη διαφάνεια ή την έλλειψη διαφάνειας ε, στη διατύπωση και λήψη αποφάσεων ε, στο πέσο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ε, συγκρού συμφερόντων, διαδικαστική δικαιοσύνη, σε δικασίες παραβάσει, ηθικά δεντολογικά ζητήματα ή και άλλα, όπως οι καζόμενες παραβιάσεις του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάποια αυτά τα θέματα μπορεί να φαίνονται απομακρυσμένα από τις καθημερινές ανησυχίες των πολιτών. Ουσιαστικά όμως που να κάνουν με το επίκεντρο της ζωής μας, με τρόπους που μπορεί να μην πάντοτε προφανής. Για παράδειγμα, μέσω του Δικτύου Ευρωπαϊκών, Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών του οποίου προεδρεύω, έχουμε ασχοληθεί με τους συναδέλφους με, σε διάφορα, με διάφορα τέτοια θέματα για να έχουμε ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και να δώσουμε αποτέλεσμα για όλου του πολίτε Ένωση. Ένα παράδειγμα είναι το πώ ε, η Frontex, ε, ο Οργανισμό Διαχείριση Εξωτερικών Συνόρων και οι διοικήσει των κρατών μελών αντιμετωπίζουν ε, αυτού που δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα ασύλου όταν του επιστρέφουν στι χώρε του. Ή με κάποιου άλλου συναδέλφου διαμεσολαβητέ είδαμε τι γίνεται με τη χρήση κάποιων ε, πιστώσεων εξαγωγών από τα κράτη-μέλη για την προστασία των ε, επενδύσεων και να δούμε αν αυτό ε, έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν για να σέβονται ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει νομίζω να αναγνωρίσουμε ότι πολλές φορές είμαστε και εμείς συνένοχοι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως εκτός ε, συνόρων. Αυτά είναι θέματα που έχουν σαφή διάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε ασχοληθεί και με άλλα θέματα, για παράδειγμα ε, την διαφάνεια του λόμπινγκ, γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν επενδυμένα συμφέροντα και η άσκηση πιέσεων έρχεται πολλές φορές σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος, ό,τι το περιβάλλον δημόσια υγεία, την ψηφιακή οικονομία και άλλα θέματα που ουσιαστικά τελικά οδηγούν και σε άρνηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι η έλλειψη διαφάνεια ό,τι αφορά τον επηρεασμό τη δημόσια πολιτική και εδώ περιλαμβάνονται στήματα όπω σύγκρουση συμφερόντων ή ε, το πέρασμα ε, από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, θα έπρεπε στον 21ο να θεωρούνται ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και αν πολύ σπάνια τα βλέπουμε από αυτό το πρίσμα. Είναι σημαντικό να δούμε, παραδείγματο χάρη, τη διασύνδεση μεταξύ τη άσκηση πιέσεων από την καπνοβιομηχανία στι Βρυξέλλε και τη συνολική επίπτωση για τη δημόσια υγεία ή τι σχέση έχουν οι πρακτικέ άσκηση πίεση και, τις, ε, και πρακτικέ τη αυτοκινητοβιομηχανία με την απόκρυψη των πολύ επιβλαβών για την υγεία εκπομπών ε, καυσαερίων στο περιβάλλον. Άρα, κακή δημόσια υγεία είναι το αποτέλεσμα. Ή τι γίνεται με του τραπεζικού μεσονομικού ε, κανονισμούς. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ε, αλληλοδιασύνδεση στον κόσμο από το 1945. Υπάρχουν αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ στις Βρυξέλλες ή στην Ουάσκτον, όμως έχουν επιπτώσεις πολλές φορές αδόκητες και απρόβλεπτες σε όλο τον κόσμο. Το 2008 αντιμετωπίστηκε ε, η κρίση, ε, μάλλον η ε, η κρίση με τις τράπεζες της ΕΠΑ οδήγησε σε κρίση και στην Ευρώπη με αποτέλεσμα μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλούς ανθρώπους αλλά έπαιξαν το ρόλο τους και οι ευρωπαϊκές τράπεζες γιατί επένδυαν στα κίνητα τα ε, αμερικανικά και βλέπουμε ακόμα τα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά αποτελέσματα επίσης βλέπουμε η ε, σημερινή αμερικανική κυβέρνηση να παίρνει πίσω κάποιες δεσμεύσεις στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και αυτό θα έχει επιπτώσει σε άλλα μέρη του κόσμου. κλιματική αλλαγή οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντο, η οργία. Πολλοί αναγκάζονται να μεταναστεύσουν και αυτό δημιουργεί κοινωνικέ και πολιτικέ πιέσει. Πολύ εμφανεί και κανεί δεν είναι στο απειρόβλητο. Μπορεί να θεωρούμε ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζει η δινή κατάσταση μια ε, αγιορική κοινότητα σε μια αναπτυσσόμενη χώρα δεν έχει και πολλά να κάνει με εμά. Ε, όταν αναγκάζεται να μεταναστεύσει λόγω τη ξηρασία που οφείλεται στην αλλαγή του κλίματο. Όταν όμω βλέπουμε τι Ανησυχίε, ανησυχίες, αναταραχές και κρατική καταστολή μπορεί να προκαλεί η σπάνιδα των πόρων και η μετανάστευση και βλέπουμε τις πολιτικές εντάσεις που δημιουργούνται και εδώ από τη μετανάστευση, τότε βλέπουμε ότι αυτός ο κύκλος είναι πλήρης. Δεν μπορεί κανείς να ε, αποδράσει από τις συνέπειες. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε αυτή την αλληλουδία σύνδεση. Μία απόφαση μπορεί να λαμβάνεται κάπου στον πλανήτη και να επηρεάζει άλλα μέρη του πλανήτη. Εμεί έχουμε διεξαγάγει έρευνες, εμπορικές συμφωνίες μεταξύ μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων χωρών του κόσμου, ώστε αυτέ οι εμπορικέ αποφάσει να μην επηρεάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ανθρώπων που ζουν πάρα πολύ μακριά από τι Βρυξέλλε. Επίση, ε, θέλουμε οι νέοι που είναι ασκούμενοι στο πλαίσιο της ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, να έχουν ίσες ευκαιρίες να πληρώνονται, να αμείβονται και να μην μείνουν πίσω από τους ήδη προνομιούχους συναδέλφους τους. Ε, επικαλούμεθα λοιπόν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και προσπαθούμε ως διαμεσολαβητές ε, να ασκήσουμε το ρόλο μας, ε, να βάλει η διοίκηση τον πολίτη στο επίκεντρο και θέλουμε να είναι ξεκάθαρα από τη μία να είναι ξεκάθαρες οι απαιτήσει του δημόσιου συμφέροντος αφενός και τα συμφέροντα των ιδιωτών αφετέρου. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το ρόλο που παίζουμε για να συνεχίσουμε να δίνουμε ζωή στην Οικουμενική Δεξιά Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, grazie. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Δώσω το λόγο στον Πατρίκ Γκασπάρ, πρόεδρο ε, του Ιδρύματος Open Society. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και όλους όσους ήρθαν εδώ σε αυτή την κοινότητα του φωτός. Χαίρομαι που εκπροσωπώ την κοινωνία των πολιτών. πραγματικά έρχομαι εδώ κατανοώντας την τιμή την οποία μου κάνετε αλλά και ε, πράγματι θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κάτι το επίγον εδώ και αυτοί που είχαν φυλακιστεί μας ζητούσαν ε, να κατανοούμε αυτά τα οποία περνούν και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτή είναι η κοινωνία των πολιτών, αυτή πρέπει να είναι. Θα πρέπει ε, αυτές τις δύσκολες εποχές να ασχολούμεθα με τα θέματα της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, όπως είχε πει η Έλενορ Ρούσβελτ Πού ξεκινούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, στα μικρά μέρη, στα σπίτια, εκεί όπου ζει ο ίδιος ο άνθρωπος, στη γειτονιά που ζει, στο σχολείο που πηγαίνει, στο πανεπιστήμιο, στο εργοστάσιο, στο αγρόκτημα, στο γραφείο. Εμείς στο Open Society, στο Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία πολιτών σε περιοχές όπως στην Σχέρα Λεόνε, ε, βοηθάμε τους νομικούς συμβούλους, βοηθάμε τους διαμαρτυρόμενους για προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Αρμενία και για αυτούς που ζητούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην Τσεχία. Ε, Εμεί προσπαθούμε να μην είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα μια αφηρημένη έννοια. Θέλουμε όμως σε αυτά τα μικρά μέρη τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, να γίνονται σεβαστά και σε πολλές χώρες που κάποτε όπως η δική μου που ήταν πρωτοπόροι για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα τώρα έχουν κάνει στροφές προς τα πίσω και πολλοί είναι ε, απογοητευμένοι από την κατάσταση αυτή. Υπάρχει ένα άγχος το οποίο ε, προσωπείται θα έλεγα από μια μείωση της έννοιας της αλληλεγγύης και την αντίληψη του ότι ε, όποιος τα καταφέρνει αυτός είναι που θα επιβιώσει. Νομίζω ότι έτσι υπονομεύουμε ουσιαστικά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό τον χώρο εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολλά όργανα που έχουν ε, λαμπρά στο παρελθόν στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι τεράστια. Απαιτείται να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές και οράματα για το μέλλον, για τους νέους, για τις νέες γενιές που πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτό απαιτεί συνεχή ε, απασχόληση και φροντίδα και δεν είναι κάτι το δεδομένο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έρθουν εδώ σήμερα γιατί τους αρνήθηκαν την βίζα ή ε, για κάποιο λόγο είναι στη φυλακή ή διώκονται γιατί εξέφρασαν την άποψή τους. 300 ε, είναι τα θύματα στον τομέα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μόνο για φέτο. Και να πω εξ ονόματος του Καβάλα στην Τουρκία, ενός πανεπιστημιακού και ο οποίος φυλακίστηκε γιατί απλά προασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως επίσης και είμαι εδώ για 13 νοτιοαφρικανούς που συνελήφθησαν εδώ και πολλά χρόνια ακριβώς γιατί προασπίστησαν το δικαίωμα του συνέχευστε και ε, της πολιτικής δραστηριότητας. Αυτά τα 70 χρόνια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ηγέτες σε περιοχές του κόσμου που δεν αντιμετωπίζουν τα δικαιώματά μας με σωστό τρόπο και ε, στις δύσκολες καταστάσεις όταν υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα τα ανθρώπινα δικαιώματα αγνοούνται. Υπάρχουν ε, ε, κάποιες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Πρώτον θα πρέπει να προασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της προάσπισης αυτών που τα προασπίζονται. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στις κυβερνήσεις που θέλουν να καταστήλουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια νέα ρητορική όπου οι κυβερνήσεις θέλουν να αποφύγουν ε, να σχολιάζονται οι καταχρήσεις τους και γι' αυτό λέγουν ότι το πρόβλημα είναι η κοινωνία των πολιτών και δήθον ονομάζουν, ονοματίζουν τα συνδικάτα, τις οργανώσεις, τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που εξαρτώνται από δυνάμεις του εξωτερικού, εχθρικές κτλ. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτές τις παγίδες. Αυτές οι αντιλήψεις μειώνουν τον αριθμό των ανθρώπων που ε, θέλουν να εκφραστούν. Ε, ο ακτιβισμός στη Ρωσία απειλείται ακριβώς γιατί δεν θέλουν οι κλεπτοκράτες ε, να ακούγονται αυτά τα οποία κάνουν. Η συζήτηση για την κοινωνία των πολιτών δυστυχώς ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά γιατί ο πρόεδρος Σορτέγκα αποφάσισε να πυροβολεί τους σπουδαστές που διαδηλώνουν και να διώκει γενικότερα τους διαδηλωτές και οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τους αντιτρομοκρατικούς νόμους ε, μόνο και μόνο για να σιωπάσουν ε, τις αντίθετες φωνές ε, και να προωθήσουν τη δική τους προπαγάνδα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προασπίσουμε όπως είπα κυρίως αυτούς ε, που παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η προσπάθεια την οποία κάνει φυσικά η κυρία Μισελ Μπασλέ και η προσωπική της ιστορία είναι καθοριστική. Όπως είχε πει και ο προκάτοχός της, ο επίτροπος Ζέντ, ε, τον Ιούνιο του 18 δεν πρέπει να είμαστε φοβισμένοι, δεν πρέπει να αποκρύβουμε από τον εαυτό μας την πραγματικότητα πρέπει να δείξουμε τι κάνουν οι άνθρωποι που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να είμαστε τολμηροί όπως είναι τολμηροί αυτοί που προασπίζονται τα δικαιώματα στην Ουγγαρία που καταγγέλουν τις επιθέσεις εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Τα δικαιώματα δεν είναι απλή ευθύνη βέβαια της κοινωνίας των πολιτών διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις όπως αυτή εδώ και οι εθνικές κυβερνήσεις φυσικά όπως και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ότι ενδιαφέρονται. Αυτό μπορεί να γίνει με τέσσερις γρήγορα το λέω τρόπος. Καταρχάς, οι αυταρχικές κυβερνήσεις ε, τη γλιτώνουν θα έλεγα διότι αποκρύβουν την πραγματικότητα, ε, δεύτερον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το ε, αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεύτερον θα πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τις ομάδες που παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι διεθνείς οργανώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την φήμη τους και το γόητρό τους για να προστατεύουν τους πολιορκημένους αυτούς μαχητές της ανθρώπινης ελευθερίας μπορούμε να το κάνουμε αυτό προσδίδοντας μια νέα θα έλεγα νομιμότητα σε αυτά τα οποία κάνουν. Δεύτερον, θα πρέπει να έχουμε ηγέτες πολιτικούς με συγκεκριμένες αρχές. Ε, υπάρχει το άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχει τους επιτρόπους τους τομείς αυτούς. Και τέλος και οι επιχειρήσεις, ο επιχειρηματικός κόσμος δεν μπορεί να αγνοεί για τα φαινόμενα διαφθοράς που υπάρχουν και βασιλεύουν στον κόσμο μας. Νομίζω ότι ε, πρέπει η κοινωνία των πολιτών να λειτουργήσει ελεύθερα υπήρξαν ιδρύματα πέρυσι τα οποία έδωσαν 40 εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις αυτές. Αλλά από την άλλη για φανταστείτε κάποιες διεθνείς επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, μεταξύ τους ο κύκλος εργασιών ξεπερνάει το 1-3. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ρόλο τον οποίο μπορούν να παίξουν. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ένα νέο όραμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα πολλές φορές τα θέματα τα δυσάριστα δεν είναι θέματα που μας αρέσει καθημερινά να αντιμετωπίζουμε. Ε, δυστυχώς παραβιάζονται και στον ψηφιακό κόσμο, εκεί όπου θα έπρεπε ε, κυρίως να κυριαρχούν οι αντίθετες αντιλήψεις. Και μάλιστα προσπάθησαν μέσα από το διαδίκτυο να δημιουργήσουν μια καρικατούρα φόβου εις βάρος του ιδρυτή μας του Τζόρτζ Σόρος και αυτές οι απειλές είναι, απειλητικές, είναι ε, αρνητικές για τη δημοκρατία και την προστασία της δημοκρατίας. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι ακριβώς η αξιοπιστία του σώματος που βρισκόμαστε σήμερα είναι υπό αμφισβήτηση. Θα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως πριν από τις εκλογές του 2019. Εδώ και δύο μήνες ζητήσατε ε, να τεθεί σε ε, υποέρευνα ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία. Θα πρέπει να απαιτήσετε από το Συμβούλιο να συνεχίσει την προσπάθεια αυτή. Και οι εκλογές του 2019 δείχνουν ότι δεν θα πρέπει να μείνετε στα λόγια και θα πρέπει ο ρόλος σας να γίνει πιο ουσιαστικός έτσι ώστε θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία δίκαιη, μια κοινωνία που να σέβεται την πολλαπλότητα και τον πλουραλισμό. Χρειάζεται να ακουστεί η φωνή μας πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα και αν θέλουμε να γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια για τα ανθρώπινα δικαιώματα τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Πρέπει λοιπόν τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν σεβαστά για ακόμη μια φορά. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι θα πρέπει κάπου να εγκαταλείψουμε το πολιτικό ρεαλισμό. Πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε κάποια λεπτά χρόνο για να ακούσουμε ερωτήσεις, να ακούσουμε παρατηρήσεις Δύο μικρές παρεμβάσεις έχουμε. Δύο παιδιών. Δύο, της Ελίζα και του Ιβάν από τη UNICEF. Να δώσω το λόγο στην Ελίζα πρώτα. Είμαι η Ελίζα από την Ιταλία. Ανησυχώ για την κατάσταση των παιδιών και των νέων στη Συρία και τη Λιβύη, όταν τα βλέπω στι ειδήσει. Πρέπει να φύγουν από τα σπίτια του, να εγκαταλείψουν τι κοινότητέ του και πολλοί από αυτού σκοτώνονται. Φαντάζομαι ότι αν ήμουν στην ίδια κατάσταση, αντιμετώπιζα εμπόλεμη κατάσταση και εγώ θα έψαχνα να ζήσω κάπου με ασφάλεια. Όπω τονίστηκε από την διακήρυξη την οικουμενική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλα τα ανθρώπινα όντα πρέπει να ζουν σε ειρήνη. Πέρα από την προέλευσή του, την καταγωγή του και αυτή είναι μια ερώτηση για την κυρία Μισελ Μπασελέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ πώς μπορούν να εξασφαλίσουν τα παιδιά που υποφέρουν θα προστατευτούν. Αυτή είναι μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Ιβάν, τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πρόσφατα διάβασα στο διαδίκτυο κάτι. Κάτι που με κλώνησε. Ένα άρθρο για την οικογενειακή βία κυρίως κατά των κοριτσιών και των γυναικών. Εξεπλάγιν. Όταν είδα ότι υπάρχει τόση βία και ότι τόσοι λίγοι άνθρωποι το ξέρουν. Παρόλο που είναι θύματα πώς θεωρούνται ένοχα τα κορίτσια. Θα είμαι ενήλικος σύντομα και θέλω την άποψή σας. Πέρα από το ρόλο σας στις διάφορες φορείς που εκπροσωπείτε, σαν άνθρωποι, τι θα κάνατε αν ξέρατε ένα κορίτσι που είναι θύμα αυτών των βιοπραγιών. Ευχαριστώ σας. Σαφέστατες ερωτήσεις. Για δύο λεπτά, όχι παραπάνω. Ε, να ακούσουμε τέσσερις-πέντε παρεμβάσεις. ΜΚΟ ή βουλευτών. Σουσκίντ. από το Βελγικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κ. Κασπάρ που μας θύμισε την κατάσταση Μαν Καβάλα που είναι στη φυλακή για ένα χρόνο. Διότι ήθελε να υποστηρίξει οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και να και έτσι βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία. Και ποια είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Χρειάζεται αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ πολυμερών οργανώσεων των κοινοβουλίων, των εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωκοινοβούλιο και οργανώσεων κοινωνιών της κοινωνίας των πολιτών. Από αυτά που είπε ο κ. Λαμπρινίδης εξεπλάγιν και όταν είπε ότι αν έχεις μάθει να μισείς, αν έχεις διδαχτεί να μισείς, μπορεί να διδαχτείς να αγαπήσεις. Αυτό άκουσα χτες ακριβώς που είχαμε έναν Παλαιστίνιο και έναν Ισραηλινό. Ο καθένας από αυτούς είχε χάσει την κόρη του από τις βιοπραγίες στην ε, Μέση Ανατολή. Και μαζί, μαζί με 600 οικογένειες στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα συμφιλίωσης. Αυτό το είπανε μπροστά σε νεολαία βελγική και αυτό είναι ένα μάθημα για το μέλλον. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Ευχαριστώ. Η Σαλίδ, Ιμπραήμ από το Κέντρο Νεολαία των Νέων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Youth Center, Youth Center for Human Rights. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή να μιλήσω Θέλω να καλέσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει πλήρω τι κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την προστασία των πασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην περιοχή μου που αντιμετωπίζονται χειρότερα από εγκληματίε, αντιμετωπίσουν κάθε είδου ενόχληση και αβάσιμες καταγγελίες, βασανιστήρια εντός που δεν ευσταθούν. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να απελευθερωθούν οι οι προασπιστές στη Μέση Ανατολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Χαντλούλ, Μπαντάουι, Αλσάντι, Βαλίντα Μπουχάιερ, Ράι Μπαντάουι, Χαμανταλινάν στη Σαουδική Αραβία, Αχμέτ Μανσούρ ε, στα Ηνωμένα Μοιράτα επίση Ραμπίρα Τζαμπ και Αμπτεχάντι Αλφαβάτ στο Μπαχρέιν και πολλούς άλλους κρατούμενους ακτιβιστές στην περιοχή κάθε ειρηνική φωνή αν κλειστεί στα κάγκελα πίσω από τα κάγκελα τότε ποιοι θα δικαιωθούν και θα ευνοηθούν οι τρομοκράτες για την κοινωνία των πολιτών δεν υπάρχει χώρος πια έχουν συρρυκνωθεί πλήρως χρειάζονται δράσεις για την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί να μην αντιδρά και μόνο όταν υπάρχουν τεράστιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη Μέση Ανατολή και στην ε, συμπεριλαμβανομένων και δολοφονιών σε πρεσβείες. Και όσον αφορά τα ανθρώπινα ε, στην Ιεμένη, είναι σημαντικό να σταματήσει ο εξοπλισμός της Σαουδικής Αραβίας. Θα συνεχίσουμε το έργο μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, των Ηνωμένων Εθνών και όλων των άλλων των θεσμών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Σιμώνα Σουριάνο από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Γεια σας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε αυτή την ημέρα και το πρωί και το απόγευμα να παρίσταμε σε μια τέτοια συνέλευση ύψης του επίπεδου με πρακτική προσέγγιση. 70 χρόνια μετά τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρισκόμαστε εδώ και ακόμα συζητούμε για το τι έγινε και πόσα μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Οι προκλήσεις είναι πάντα και ε, πιο επικίνδυνε σε ένα ψηφιοποιημένο, παγκοσμιοποιημένο κόσμο και ε, καμιά φορά είναι δύσκολε οι αρχέ που παρουσιάζονται. Δύσκολο να βρει κανεί τα όρια μεταξύ εκείνου που είναι σωστό και αυτού που είναι λάθο. Η Ιταλία θε, έχει κάνει διάφορες, ε, θέλει να προσπαθεί να, προλάβει την καταπίεση και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μα εστιάστηκε ιδιαίτερα στα τρόπινα δικαιώματα και ξεκινήσαμε διάφορε έρευνε για να συλλέξουμε στοιχεία όσον αφορά την ισοτιμία των φύλων, όσον αφορά τη βία κατά θρησκευτικών μειονοτήτων. Ε, Επίση, όσον αφορά το διεθνέ εμπόριο, να μην λησμονούμε ότι καμιά φορά το άνοιγμα στο διεθνέ εμπόριο μπορεί να προκαλέσει αλλαγές όσον αφορά τους κανόνες στην εθνική νομοθεσία και έτσι να τροποποιηθούν τα κοινωνικά και αστικά δικαιώματα. Μετά εγώ θα, θα ήθελα να υπάρχει μια επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και θα ήθελα ότι εξελέγει εντός του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Ιταλία ε, ομόφωνα για την προστασία και την πρόληψη τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να γίνει αυτό χρειάζονται πολλέ παρεμβάσει. Μόνο, όχι μόνο ειδικέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρεμβάσει, αλλά και άλλε ε, στον τομέα, το, το αναστικό, ε, στο σύστημα προόνοια, για την εργασία. Πρέπει να γίνεται καλύτερη κατανομή του πλούτου, ώστε να ξεπεραστεί η απόλυτη φτώχεια από την οποία πλήττεται ακόμα δυστυχώ η Ιταλία. Θα θέλαμε να υπάρχει αξιοπρεπής είσοδος στην αγορά εργασίας, να υπάρχει μια παιδεία εγγυημένη που θα παρέχεται σε όλους και αυτά είναι κάποια μέτρα τα οποία θεσπίζουμε όπως η καταπολέμηση τη συγκρούσεων συμφερόντων. Είναι μέτρα όλα αυτά που κατά την άποψή μου κινούνται προς την κατεύθυνση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνουμε σημαντικά βήματα όσον αφορά την επιβεβαίωση κάποιων αρχών των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά είναι σαφές ότι ο δρόμο και οι προκλήσει γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και γι' αυτό πιστεύω ότι και μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με έναν τρόπο αποφασιστικό και συγκεκριμένο για τα κοινωνικά και, αστικά και πολιτικά δικαιώματα που θα πρέπει να παγιωθούν στην Ευρώπη δεν μπορεί παρά να βοηθήσει την Ιταλία και τα κράτη-μέλη προφανώς να προωθήσουν και να υπερασπιστούν αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα, Ραφαέλ Σανουή Αλζάν από, τον Οργανισμό κατά της α, ε, θανατικής ποινής. Ευχαριστώ πολύ. Διεθνής Οργάνωση κατά της θανατικής ποινής. Θα ήθελα να αναφερθώ στην διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι σημαίνει για τον κόσμο σήμερα. Δύο βασικά είναι τα σημεία στα οποία εγώ πιστεύω ότι έχει πολλά προσφέρει η διακήρυξη αυτή. Καταρχάς, η προσπάθεια να έρθουν σε ένα κοινό επίπεδο οι τρόποι προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεύτερον η έννοια του καθολικού χαρακτήρα. Το άρθρο 3 της διακήρυξης λέει ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια. Αυτό το δικαίωμα στη ζωή στο άρθρο 3 είναι θα έλεγα το σημείο εκκίνησης ε, τις προσπάθειες που κάνουμε σε όλο τον κόσμο για την κατάργηση της θανατικής ποινή. Μετά υπήρξε και το Διεθνές ε, ε, Ποινικό Δικαστήριο. Υπήρξαν τα πρωτόκολλα 6 και 13 υπήρξε και η σύμβαση της Αμερικής όπως λέγεται και πολλά άλλα πρωτόκολλα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω πάντως τη σημασία του καθολικού χαρακτήρα ε, στην καταπολέμηση της θανατικής ποινή και στην προώθηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις 10 Οκτωβρίου είχα πάει στην Κίνα με πολλούς άλλους δικηγόρους και διανοούμενους και συναντηθήκαμε με συζύγους πολιτικών ε, κρατουμένων Όλοι μου είπαν ένα πράγμα, όλοι μου ζήτησαν να πω ότι μην επιτρέψετε στις κινέζικες αρχές να προωθούν την ρητορική τους στην, για τα ανθρώπινα δικαιώματα λέγοντας ότι κάθε χώρα έχει τα δικά της επίπεδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι. Λοιπόν, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικού χαρακτήρα. Το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην κατάργηση της θανατικής ποινής, την ελεύθερη έκφραση, ε, τα δικαιώματα ακόμα και των κρατουμένων. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι τα ίδια στον κόσμο. Ε, στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, στην Κίνα, στις Ηνωμένε Πολιτείε ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το δικαίωμα στη ζωή επίσης. Έχει υπάρξει τις τελευταίες δεκαετίες πρόοδο στον τομέα της κατάργησης της θανατικής ποινή Πάνω από τα δύο τρίτα των μελών των Ηνωμένων Εθνών είτε έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή είτε δεν την εφαρμόζουν. Τον, στις 27 Φεβρουαρίου ε, του 19 σε αυτήν εδώ την αίθουσα θα υπάρξει εναρκτήρια ε, συνεδρίαση του Παγκόσμιου Κογκρέσου για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Ε, θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους να έρθετε σε αυτό το Κογκρέσο το Διεθνές για να ξεκινήσει ο διάλογος για τη μελλοντική στρατηγική στον τομέα των προσπαθειών κατάργησης. Ε, το οφείλουμε αυτό στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βουλευτές, ε, οι ευρωβουλευτές, οι εθνικοί βουλευτές, οι διπλωμάτες ε, και η κοινωνία των πολιτών. Ε, η συνάντηση αυτή θα οργανωθεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Βελγίου, της Ελβετίας και, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα τελειώσω και εγώ με κάτι είπε ο, ο Μαντέλα θα έλεγα δεν είναι απλά μια αναφορά στο Μαντέλα. Ε, είπε ότι η θανατική ποινή είναι μια βαρβαρότητα, είναι μια επιβίωση του ενστίκτου του ζωικού στα ανθρώπινα όντα σήμερα. Ένα λεπτό, Μάνφρετ Νόβακ. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε ότι το κράτος δικαίου, η δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα παντού στον κόσμο αντιμετωπίζουν ε, μια πάρα πολύ βαθιά κρίση με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την ε, ε, οικουμενική διακήρυξη ως τη μεγαλύτερη. Και λόγος είναι οι μεγάλες ανισότητες που αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε και αυτά προσκάπτουν την κοινωνική συνοχή και το δημοκρατικό ιστό των κοινωνιών μας οδηγώντας την ριζοσπαστικοποίηση, των εξτρεμισμών και τη βία. Πρέπει λοιπόν να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν αντιμετωπιστούν ε, τα αίτια της πολλαπλής κρίσης που βιώνουμε σήμερα. Χρειάζεται δηλαδή μία αναστροφή σε ό,τι αφορά την οικονομική και κοινωνική πολιτική της Ένωσης, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα δράση τη Βιέννη και την οικονομική διακήρυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός πολιτικός πολιτικό-οικονομικό πρωταγωνιστής. Μπορεί να ηγηθεί με το παράδειγμά τη αυτή την αναστροφή. Αυτό περιμένουν ε, οι εκατομμύρια υπερασπιστών δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο. Να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα έχουμε κοινέ αξίε, αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και θα σα δώσω δύο σύντομα παραδείγματα. Το πρώτο, το αδιέρετο, η ισότητα, η αλεξάρτηση ε, των ανθρώπινων όντων είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρότητα και να προωθήσουμε ε, αυτά τα δικαιώματα όπως τα πολιτικά και τα αστικά. Και δεν θέλουμε να περιστήλουμε το κράτος πρόνοιας. Αντίθετα να μειώσουμε τις ανισότητες, να προωθήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή είναι η στόχη. Δεύτερον, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο ώστε να υπάρχει ευαισθητοποίηση στις αξίες, ε, στα άπρα δικαιώματα, τη δημοκρατία, στο μυαλό, ε, σε αυτούς που νιώθουν ότι έχουν μείνει πίσω, για να δημιουργήσουν περισσότερη αγάπη, όπως είπε και ο Σταύρος. Ε, την αγωγή του πολίτη πρέπει να προωθήσουμε. Έχουμε το στόχο θεμελιώσιμης ανάπτυξης 4 και από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο πρέπει να εμφυσίσουμε αυτές τις αξίες. Το Παγκόσμιο Κάμψο των Δικαιωμάτων είναι έτοιμο και θα είναι ένας ισχυρός εταίρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε περισσότερε πλέον δραστηριότητε στον τομέα τη αγωγή των πολιτών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Well, thank you so much, uh, Mr. Michel, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ελίσα μου έκανε ένα ερώτημα ε, προσωπικό. Τι μπορούμε να κάνουμε για την προστασία των παιδιών. Φυσικά δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το δικό μου γραφείο εγώ είμαι και παιδίατρος, ξέρετε. Δεν είμαι μόνο μητέρα και γιαγιά, είμαι και παιδίατρος. Και όπου πάω και όπου θα πάω και στο μέλλον θα μιλώ πάντοτε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών. Γιατί εδώ και χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Αυτό πρέπει να γίνει σε πολλά επίπεδα. Στο ε, κυβερνητικό πρέπει να βοηθήσουμε κυβερνήσεις να κάνουν το σωστό, να επενδύσουν στα παιδιά. Και έτσι ε, δίνοντάς τους δηλαδή παιδεία, περίθαλψη, από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Αυτό θα εξασφαλίσει στη χώρα το μέλλον της. Τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύουμε, να τα ταΐζουμε, να τα στηρίζουμε. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε πολύ από πολιτικής πλευράς, κοινωνικής πλευράς και στις γυναίκες, διότι οι γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντικές όχι ότι και οι πατεράδε δεν έχουν ευθύνη, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Απλά λέω ότι πρέπει να χειραφετηθούν οι γυναίκε, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό παράγοντα τη κοινωνία για την προστασία των παιδιών. Και εγώ προσωπικά εργάστηκα με τη UNICEF και με άλλου συναδέλφου για να δημιουργήσουμε συνέργειε, εταιρικέ σχέσει για τη σωστή σύστημα των Υπάρχει η λέξη της ε, ε, καθοδήγησης, της δημιουργίας δυνατοτήτων, ε, ε της τεχνικής συνεργασίας, ιδίως σε θέματα δικυβέρνησης κράτους δικαίου. Υπάρχει το λεγόμενο advocacy, αλλά έχουμε και ένα σημαντικό στόχο, υποχρέωση να προωθήσουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Να δημιουργήσουμε συνέργειες ε, με άλλους για να το πετύχουμε αυτό. Είναι σημαντικό. Θα μπορούσα να μιλάω και για ώρες βέβαια, γιατί με παθιάζει το θέμα αυτό. Πρέπει το θεματολόγιο 2030, στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να ε, τους πετύχουμε αυτούς τους στόχους και στο Κατοβίτσε της Πολωνίας ε, η διάσκεψη των συμβαλωμένων μερών, η COP24, ε, πρέπει να πετύχει. Γιατί αν δεν αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, δεν θα έχουμε δικαιώματα. Ούτε για τα παιδιά, ούτε για τι μελλοντικέ γενιέ. Και οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη και όλοι οι άλλοι στόχοι που πρέπει να περιλαμβάνουν πάντοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να φροντίσω να μην μείνει πίσω κανένα παιδί. Εγώ θα υψώνω τη φωνή μου και στη συνέχεια και θα κάνω ό,τι μπορώ για να το εξασφαλίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Κλοντ Μωράες, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Για το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνιο. Θα φορούσα τα ακουστικά μου, αλλά τόσα λίγα Ιταλικά τα καταλαβαίνω. Αντώνιο, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω ασυνήθιστο καθήκον. Είναι σκοτσέζικη η προφορά μου, ε, αν διερωτάστε τι προφορά έχω. Ναι, λόγω μετάφρασης καθυστέρησε το γέλιο. Ε, λόγω διερμηνίας. Να εξηγήσω, να εξηγήσω στο Μισελ Μπασελέ. Μισελ, κάτσε μισό λεπτό να σου εξηγήσω. Γιατί είμαι Σκοτσέζο. Γιατί είμαι Σκοτσέζο. Να σου πω κάτι. Ε, ξύπνησα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαι ειδική καταγωγή. Αλλά σαν παιδί θα μαντεύει τι γίνεται όσο εξηγώ. Ευαισθητοποιήθηκα τη δεκαετία του 70, το 78. Ο αδερφός μου και εγώ καθόμαστε στο σπίτι και ξαφνικά οι γονεί μου λένε Ζούσαμε στο Στέρλινγκ, στη Σκοτία. Θα ξέρεις θέλω να πω. Και λέει δυστυχώ: θα έχουμε κάποιους που θα μείνουν μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πανεπιστημιακοί, δεν σε καλή κατάσταση. Ξέρεις τι θα πω. Έχουν παιδιά. Τα παιδιά ε, είναι, έχουν βασανιστεί, είναι χάλια. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Και στα παιδιά είχαμε μεγαλύτερο σπίτι. Είχαμε τότε χιλιανούς πρόσφυγες και μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τι είναι το βασανιστήριο. Το 1978 τα παιδιά μου εξήγησαν τι είναι τα βασανιστήρια. Και τότε κατάλαβα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ένα χρόνο αργότερα η κυρία Αλιέντε είδε στην πόλη μας και μου έδωσε μια φύσα που έχω στο γραφείο μου πάνω. Εκεί ευχαριστεί τον πληθυσμό της πόλης που υποδέχτηκε αυτό που τώρα γνωρίζουμε ότι είναι πρόσφυγες προσφύγες από την Χιλή τη δεκαετία του 70. Πριν φύγεις, είσαι από τη Χιλή, δεν σε είχα συναντήσει, αλλά νομίζω ότι σε ξέρω, γιατί νομίζω ότι ξέρω τι ήταν οι χιλιανοί πρόσφυγες. Έτσι ευαισθητοποιήθηκα για τους πρόσφυγες. Δεν τα είχα γράψει αυτά, δεν ήταν κανονικά συμπεράσματα. Όταν σε είδε θα σου εξηγήσω. Και αν κάποιο σου πει ότι δεν καταλαβαίνει, κάποιο άλλο δεν καταλαβαίνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, εσύ ξέρω ότι τα καταλαβαίνει. Ευχαριστώ πολύ για τα πάντα. Λοιπόν, θα αναφέρω το Σταύρο Λαμπρινίδη. Άργησα και άργησα γιατί ο Αντώνιο είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο και η Επιτροπή μα ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πει κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω θα πηγαίνει καλούτσικα. Είμαστε σε μια ακρόαση τώρα για την Πολωνία. Η Πολωνία έχει προβλήματα με το δικαστικό τομέα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην Ουγγαρία. Σε πολλά κράτη-μέλη καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Όταν ακούσα το Σταύρο Λαμπρινίδη, που είναι ο εκπρόσωπος για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση στον υπόλοιπο κόσμο, θα συμφωνεί με αυτό που θα πω τώρα Αντώνιο. Πρέπει να συσχετίσουμε τις δικές μας αξίες και να μην θεωρήσουμε δεδομένα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε τα του οίκου μας εντάξει πριν αρχίσουμε να κηρύττουμε σε άλλε χώρε τι να κάνουν ή υπογράφουμε συμφωνίες και συνεργαζόμαστε με κράτη άλλων περιοχών του κόσμου. Να είναι ξεκάθαρο στο κρατήριο αυτό που πολεμάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μίλησε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ο σταύρο. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε ημέν με τους δε αν δεν έχουμε τον ίδιο σεβασμό για την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κλείνοντας πάνω σε αυτό. Ο Πάτρικ από το Open Society Institute αναφέρθηκε στην Eleanor ε, Roosevelt. Και όλα ξεκινάνε με τα άτομα, κοντά στο σπίτι σου τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν δύο προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα που διαφαίνονται. Το πρώτο, και γι' αυτό είσαστε εδώ, και γι' αυτό συγκαλέσαμε τη συνεδρίαση, για την οποία ευχαριστώ την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον πρόεδρο γι' αυτό. Έλεγα λοιπόν, το συζητάμε, διότι είτε τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται κάτι πολύ αόριστο και πολύ ευρύ σαν έννοια, άρα τα πάντα είναι ανθρώπινα δικαιώματα και αγνοούμε το θέμα, ή είναι παντού τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μάχη δίνεται παντού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πριν έρθω στην ε, Σκοτία, γεννήθηκα στην Ιεμένη. Όταν κάποιο ανέφερε ε, την Ιεμένη, εγώ γεννήθηκα στο Άντεν και με τον πόλεμο ε, απελάθηκα. Και είχαν διαπραχθεί φρικαλότητε τότε, αλλά ήμουν πολύ μικρό για να καταλάβω και να θυμάμαι. Η, η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τεραστίου μεγέθου σε όλο τον κόσμο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωση ε, μας τα παρουσιάζουν κάθε μέρα στα σπίτια μας. Συντομότατο το συμπέρασμα μου εγκατακλείδη. Τι θέλω να πω Αντώνιο, ότι σήμερα αν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση των Αξιών πρέπει να ερμηνεύσουμε τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν κάτι που θα πρέπει να ανανεωθεί, να, ανανεωθεί, εξυγχρονιστεί και ότι να δούμε ότι είναι κάτι που έχει πρακτικές εφαρμογές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που μας δένει όλους μαζί, μας δεσμεύει. Οι πρόσφυγες στο στρατόπεδο της Μόριας στην ε, Ελλάδα ή στο Αργαντέ στον Ήγυρα, οι πρόσφυγες ε, που είναι σε κέντρα κράτησης στη Λιβύη που τους είδα και βασανίζονται και επιστρέφονται παρόλα αυτά στους τόπους από όπου ήρθαν και τελικά αυτοί αυτοκτονούν σε μεγάλα ποσοστά και πεθαίνουν και δεν θέλουν να επιστρέψουν. Είναι όλοι άνθρωποι όλους τους καλύπτει η καθολική διακήρυξη των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και πρέπει να βρούμε εμεί τι λύσει, να πολεμήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου αυτά υπάρχουν. Καλό που συνεκλήθη μια τέτοια σημαντική συνεδρίαση που συμμετέχουν τόσο σημαντικοί άνθρωποι που πολεμούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκπροσώποι τη κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ. Πολλοί από εσά ξέρετε πολλά περισσότερα από εμά, από πολλού από εμά. Θέλω να σα ευχαριστήσω όταν είσαστε πολύ, είσαστε όλοι πολύ κουρασμένοι, δουλεύετε όλη μέρα, ήσασταν το πρωί στις συνεδριάσεις, ξεκινήσατε εδώ στις 3, άρα είχα το άσχημο καθήκον να έρθω τελευταίος, τελευταίος και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους όλους διοργανωτές. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να πολεμάει κάνεις ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι που είναι πιο ρεαλιστικό, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το προωθούμε καθημερινά. Αυτό έκαναν οι μιλητέ σήμερα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω απ' όλα για τη συμμετοχή σα και εκ μέρου όλων των συναδέλφων και ευχαριστώ Αντώνιο για αυτή την ευκαιρία που μας δόθηκε. Ελπίζω να απολαύσετε τις σημερινές εργασίες και να πήρατε και κάτι από το σήμερα. Αυτή η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να γίνει ένα εργό σημαντικό έγγραφο, όχι ένα κομμάτι χαρτί, αλλά κάτι για το οποίο να πολεμάμε καθημερινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια μέρα που δεν ολοκληρώθηκε ακόμα, διότι ετοιμάζουμε το δεύτερο πάνελ. Και εν αναμονή του δεύτερου πάνελ θα δούμε βίντεο με μαρτυρίες διαφόρων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ αυτούς που συμμετείχαν στο πρώτο πάνελ. No effort for humanity is in vain.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 ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo mrežu romskih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 aktivnostima odem u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća, najveća povratna informacija i kad vidim i kad osetim da ih mu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 kontakter. Yeah. So, ladies and gentlemen, may I please ask you now to be um, seated. Παρακαλώ καθίστε κυρίες και κύριοι. σωστό. Λέγομαι David McAllister. Είμαι ευρωβουλευτής ε, και έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και έχω την τιμή και σήμερα να προεδρεύω του δεύτερου πάνελ αυτής της διάσκεψης ε, με θέμα τους ε, μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μπορείτε να το έχετε ξανακούσει εδώ στις Βρυξέλλες ότι είναι μια πάρα πολύ βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λέει και το άρθρο 2 της Ένδειξης Λισαβόνας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίω στο Ευρωκοινοβούλιο που ηγείται και τιμά θαραλέους ανθρώπους και οργανώσεις που προωθούν, υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δίνουμε το βραβείο Ζαχάροφ, το οποίο το πρωταπονήμα πριν από 30 χρόνια. Πέντε βραβευθέντες πήραν και το βραβείο Νομπέλ, μεταξύ αυτών και το 18. Νάντια Μωράτ και Ντένις Μουκβέγγε πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σα είπα ότι είμαι και γνωρίζω πολύ καλά πόσο σοβαρά ε, λαμβάνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και εντό και εκτό ευρωπαϊκών συνόρων και τη σχετική μα δέσμευση. Καταθέτουμε ψηφίσματα, διενεργούμε επίσημε επισκέψει Έχουμε συναντήσει των αντιπροσωπιών μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια και επίσης εκλογικές, ε, επιτροπές εκλογικής παρατήρησης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει αλματώδη βήματα για να προωθήσει σε παγκόσμιο επίπεδο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά γνωρίζουμε σίγουρα ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν. Η πρόληψη, η ταχεία αντίδραση πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να λογοδοτήσουν αυτοί που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουν παγκόσμιου μηχανισμού, θέλουμε ψηφιακέ, τεχνολογικέ αλλαγέ να μην είναι σε βάρος ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η 70η επέτειο από την υιοθέτηση τη Οικουμενική Διακήρυξη είναι σίγουρα μια αφορμή να γιορτάσουμε, αλλά να προβληματιστούμε για το τι θα πρέπει να γίνει και στο μέλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση με διεθνούς, διεθνείς ηγέτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ολόκληρο τον κόσμο. Καλωσορίζω του πέντε προσκεκλημένου μα εδώ στο πάνελ, οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί μας ε, την εμπειρία του για το πώ μπορούμε να προωθήσουμε την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δικαιωμάτων σε έναν κόσμο μεγάλε προκλήσει. Θα συζητήσουμε τι συνέργειε, το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία για την πρόσθεση του διεθνού ε, δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώ θα προωθήσουμε του διεθνεί περιφερειακού μηχανισμού. Όλοι οι ομιλητέ το γνωρίζουν, αλλά θα τους παρακαλέσω να τηρήσουν ε, το δεκάλεπτο που έχουν στη τους. Πρώτος ε, ο κύριος Τόρμπον Γιάκλαντ, γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δυστυχώς όμως δεν μπορεί να είναι μαζί μας ε, εδώ διαζώσεις. Όμως θα μας... θα δούμε ένα μήνυμα που έχει στείλει. Έπειτα θα λάβει το λόγο ο κύριος ε, Ερνάντεφ Καρσία από την Διαμερικανική Επιτροπή, ε, Γκόι Λούμπου από την ε, Αφρικανική Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Δικαιωμάτων των Προσώπων, Καταρίνα Γκάρντα Χφάτζε πρώτη αναπληρώτρια διευθυντή ε, του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, της ΟΑΣΕ. Μπεάτε Ρούντολφ επίση, θα μας μιλήσει, πρόεδρος τη Global Alliance of National Human Rights Institutions και μέλος ε, του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Αντίστοιχου Δικτύου, κάθεται δίπλα στον κύριο Λούμπου και θα ολοκληρώσει η καθηγήτρια Πάμελα Πάλματερ, που είναι δικηγόρος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ράισον του Τορόντο, του Καναδά. Επίσης θα έχουμε και μία συνεδρία αποκρίσεων. οποίο θέλει το λόγο θα ήθελα να το παρακαλέσω να συμπληρώσει το έγγραφο που έχει στο φάκελο του και να το στώσει σε κάποιον κλητήρα. Αυτά από πλευρά μου και θα ξεκινήσουμε ακούγοντα πρώτα την προσφώνηση του Θόρμπρον Γιάγκλαντ με ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθότι γιορτάζουμε την 70η επέτειο τη Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και για πρώτη φορά ορίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται στον πλανήτη μα. Δύο χρόνια μετά, το Συμβούλιο τη Ευρώπη εγκρίνει την Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ένα μοναδικό για όλη την Ήπειρο ε, συλλογικό σύστημα σύστημα το οποίο εγγυάται δια νόμου τα δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνει η Οικουμενική Διακήρυξη και τα οποία εφαρμόζονται με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδράζει στο Στρασβούργο. Η σύμβαση αυτή αλλά και οι επόμενες συνθήκες μετασχημάτισαν την Ευρώπη, τη μεταμόρφωσαν σε κάτι καλύτερο. Έχουμε ίσια δικαιώματα για τα παιδιά, ε, είτε γεννιούνται εντό είτε εκτός γάμου, από ποινικοποίηση των ε, ομοφυλόφιλων ε, ζευγαριών. Είναι η κατάργηση επίση επίσης ε, της θανατική στην Ευρώπη είναι σημαντικό. Και αυτά δεν έγιναν έτσι τυχαία. Έγιναν λόγω του ότι ε, ρίζωσε εδώ ε, μια κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζεται από την σχετική νομοθεσία. Είμαστε περήφανοι σήμερα που μπορούμε να συνεργαζόμαστε με πολυμερείς εταίρου μεταξύ των οποίων την Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία έχουμε μια ειδική εταιρική σχέση. Πολλέ φορέ η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη Ευρώπη ω βάση για τη δράση τη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Και το Συμβούλιο τη Ευρώπη ε, από την πλευρά του ε, υλοποιεί πολλά έργα με βάση τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρούμε ε, και προσπαθούμε να προωθήσουμε τι κοινέ μα αξίε στην επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Όμω σήμερα στην Ευρώπη βλέπουμε την άνοδο του ακραίου εθνικισμού και λαϊκισμού. Αυτά υπονομεύουν το πολυμερή χαρακτήρα, του θεσμού μα, τις πολύ σημαντικέ κοινέ αξίες που μας ενώνουν. Αυτή λοιπόν η Εβδομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να γίνει ευκαιρία. Όχι μόνο για να τονίσουμε τη συνεργασία μας, αλλά ε, και θέλω να πω ότι μιλάμε για συνεργασία με κυβέρνηση και με την ε, κοινωνία των ε, πολιτών, αλλά επαναλαμβάνω να υψώσουμε τη φωνή μα και με περηφάνεια να μιλήσουμε για τα όσα έχουν πετύχει τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλου του Ευρωπαίου ε, στα κράτη-μέλη. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να πάει προ τα εμπρό και όχι προ τα πίσω. Εύχομαι λοιπόν μια επικοδομητική εβδομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλέ εργασίε στη διάσκεψή σα. Okay, was... Ωραία. Ο κύριος Γιάνκμαν έστειλε αυτό το τηλεμήνυμα. Ο κύριος Ζωέλ Χερνάντες Καρσία έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μακάλιστερ, αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι. Η Αμερικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Χαίρετε που είναι εδώ για την επέτειο, την 70η της ε, διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακαλώ να δεχτείτε την αναγνώριση της Διαμερικανικής Επιτροπής για το έργο που επιτελεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα εορτάζουμε την 70η επέτειο ε, της καθολικής αυτής διακήρυξης. Στην Αμερικανική Ήπειρο εορτάζουμε επίσης την 70η επέτειο τη ιδρύσεως της οργάνωσης των Αμερικανικών ε, κρατών και τη έγκριση τη αμερικανική διακήρυξη Δικαιωμάτων και Καθηκόντων του Ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 χρόνων, το καθολικό και διαμερικανικό σύστημα προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων λειτουργούσαν παράλληλα και τώρα αλληλοενισχύονται. Το περιφερειακό σύστημα τροφοδοτήθηκε από οδιαγραφέ και τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν στην Ηνωμένα Έθνη. Το διαμερικανικό σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένα προϊόν σταδιακής εξέλιξη του συστήματος η διάσκεψη του Τεπέκ ήταν ακρογωνίως λίθος, ήταν καμπή μάλλον στην διοργάνωση αυτού του ημισφαιρίου και διεφάνισαν τότε ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ετοιμασία για τη διάσκεψη του Σαν Φρανσίσκο, η κυβέρνηση του Μεξικού ε, συνεκάλεσε την διαμερικανική διάσκεψη για τα προβλήματα του πολέμου και τη ειρήνης που έγινε στο Τεπέκ από 21 Φεβρουαρίου με μέχρι 8 Μαρτίου 45, 1945. Σκοπός ήταν οι κυβερνήσεις των Αμερικανικών χωρών της Αμερικανικής Υπήρου να εξετάσουν από κοινού τη συμμετοχή της Αμερικής στη μελλοντική οργάνωση. Όσο αφορά ε, το, ψήφισμα που αφορούσε την διεθνή προστασία των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου, η διάσκεψη επέλυσε με αυτόν τον τρόπο να αναθέσει στην Διαμερικανική Δικαστική Επιτροπή τη σύνταξη ε, προλίου, πρωτολίου διακήρυξη των διεθνών δικαιωμάτων και καθηκόντων του ανθρώπου που θα έπρεπε να θετηθεί από τη μορφή τη σύμβαση. Θα, αργότερα θα ενέκρινε την Αμερικανική Διακήρυξη και Αμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το ε, αμερικανικό σύστημα εξελίχθηκε τάχιστα το, με το τέλο ε, του Δευτέρου ε, Παγκοσμίου Πολέμου, τη στιγμή που η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών ενεργοποιήθηκε. 25 ε, κράτη τη Αμερικανική Υπηρείου συναντήθηκαν στην Ποκοτά τη Κολομβία τον Απρίλιο του 1948 και οθέτησαν τη χάρτα τη οργάνωση των Αμερικανικών κρατών, την Αμερικανική συνθήκη των λύσεων του Ειρηνικού και την Αμερικανική διακήρυξη του δικαιωμάτων και καθηκόντων του ανθρώπου. Η Αμερικανική διακήρυξη υιοθετήθηκε μήνε πριν από την Καθολική διακήρυξη και υπογράμμισε τη δέσμευση τη περιοχή για διεθνή προστασία των ανθρωπίνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικοδοποίησε ένα βασικό κατάλογο αστικών, πολιτικών και οικονομικών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, η Αμερικανική διακήρυξη εμπεριέχει μια σειρά καθηκόντων για το λαό. Η Αμερικανική διακήρυξη είναι διαφορετική από το δόγμα μέσω του οποίου το κράτος χορηγεί δικαιώματα στους πολίτες αυτού και ακολουθεί το δόγμα, το, το φυσικό νόμο των δικαιωμάτων που είναι εγγενή των ανθρωπινών. Η πρώτη παράγραφος του προημίου λέει όλοι οι άνθρωποι γεννούνται ελεύθεροι και ε, ισότιμοι, έχουν δικαιώματα ε, και αξιοπρέπεια και πρέπει ε, τις έχουν επίγνωση από τη φύση, πληκισμένοι με επίγνωση. Γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν σαν αδέρφια το ένα το άλλο. Αναγνώρισαν τα Αμερικανικά κράτη ότι όταν το κράτο νομοθετεί επ' αυτών δεν χορηγεί δικαιώματα, αλλά αναγνωρίζει δικαιώματα τα οποία υπάρχουν ανεξάρτητα από τη δημιουργία ενό κράτου. Η ιδέα ενό νομικά δεσμευτικού μέσου ανανεώθηκε στη διαβούλευση των Υπουργών Εξωτερικών στο Σαντιάγο τη Χιλής τον Αύγουστο του 1959. Οι Υπουργοί Εξωτερικών υιοθέτησαν ένα ψήφισμα με δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα ανέθεσαν στο Διαμερικανικό Συμβούλιο των Δικαστών να συντάξουν μια σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με θεσμού για την εφαρμογή των δικαιωμάτων. Άλλη πλευρά ενέκριναν τη δημιουργία Διαμερικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για να πετύχουν του στόχου τη μελλοντική συμβάσεω. Η επεξεργασία τη Αμερικανική Σύμβαση χρειάστηκε 10 χρόνια. Η διαδικασία σταμάτησε ενώ το Διεθνέ Σύμφωνο για Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνέ Σύμφωνο για Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα υιοθετήκε τι 16 Δεκεμβρίου του 1966 και αυτά ήταν μα. Με διαπραγμάτευση εντό του ΙΕ. Η Οργάνωση Αμερικανικών Κρατών εξέτασε τη συμβατότητα μεταξύ των καθολικών αυτών εργαλείων και αυτού του, για, το εργαλείο για το ημισφαίριο συμπεραίνοντα ότι η Αμερικανική Σύμβαση θα έπρεπε να προσεγγίσει το θέμα από περιφερειακή πτωχή. Αργότερα η Αμερικανική Ειδική Διάσκεψη της, για ανθρώπινα δικαιώματα στο Σαν Χωζέ τη Κωνσταντίνα θέτει την Αμερικανική Σύμβαση στι 22 Νοεμβρίου του 1969. Το σύμφωνο του Σαν Χωσέ ετέθησε ισχύ στις 18 Ιουλίου του 1978 όταν επετέθησαν 11 αναγκαίες κυρώσεις, επικυρώσεις. Η Αμερικανική Σύμβαση στο πρώτο τμήμα καθορίζει τα, τα ε, καθήκοντα των κρατών και τα δικαιώματα των ατόμων. Στο δεύτερο τμήμα, η Αμερικανική Σύμβαση καθορίζει του τρόπου προστασία. Η Διαμερικανική Επιτροπή και το Διαμερικανικό Δικαστήριο, που είναι αρμόδιο φορεί για να εξετάσουν υποθέσει που αφορούν τη συμμόρφωση με τι δεσμεύσει που αναλάβουν τα συμβαλώμενα μέρη τη Συμβάσεω. Το διαμερικανικό σύστημα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτίζεται από δύο φορεί, την Διαμερικανική Επιτροπή και το Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή είναι βασικό φορέα οργανώσεω Αμερικανικών κρατών, αλλά το Δικαστήριο είναι ένα φορέα στι συνθήκε που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου τη Αμερικανική Σύμβαση. Το Αμερικανικό σύστημα ενεπνεύστη από το αρχικό ευρωπαϊκό σύστημα. Η Αμερικανική Ήπειρο διατήρησε του δύο θεσμικού μηχανισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει πρωτόδικα τι υποθέσει. Αν δεν διορθωθούν ε, οι παραβιάσει σε αυτό το επίπεδο, μπορεί η Επιτροπή να μηνύσει το κράτος και να το προσάγει στο δικαστήριο. Και αποφάσεις του δικαστηρίου είναι τελεσίδικες και δεσμευτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ε, εντολή απορρέει από τη μαρική διακήρυξη των δικαιωμάτων και καθηκόντων του ανθρώπου, την Αμερικανική Σύμβαση, η Επιτροπή βασίζεται σε τρει πυλώνε: στο σύστημα αναφορών και υποθέσεων, η εποπτεία τη καταστάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αμερικανική Ήπειρο και το πρόγραμμα τεχνική συνεργασία. Έχει μοναδική εντολή. Αυτό ο φορέα απαρτίζεται από 7 επιτρόπου και επικουρείται από εκτελεστική γραμματεία και έχει αρμοδιότητα πάνω στα 35 κράτη-μέλη τη Οργανώσεω Αμερικανικών Κρατών και μέσω τη θεματική αναθέσεω εκθέσεων που δικαιώματα δικαιωμάτων των γυναικών, μεταναστευτών, των παιδιών, των εφήβων, των ηθαγενών πληθυσμών, του πρασπιστέ των, των ε, ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ΛΟΑΔ και ανθρώπου που έχουν στερηθεί τη ελευθερία του. Ε, και επιπλέον έχει δύο ειδικέ ε, δυνατότητε για εκθέσει για την ελευθερία τη έκφραση, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και δικαιώματα. Μέσω αυτού του συστήματο παίζει η ρόλο δικαστηρίου. Η Επιτροπή ε, λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να προστατεύσει τη ζωή και κεραιότητα ανθρώπων σε κίνδυνο. Πέραν αυτών, ακούει καταγγελίε για παραβιώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προστατεύονται από μέσα που είναι πηγέ ε, τη εντολή τη Επιτροπή. Η Επιτροπή επίση απολαμβάνει συμφιλωτικέ εξουσίε για να επιλύσει ε, με φιλικό τρόπο διάφορε υποθέσει. Το ρασιόνε περσόνα τη Επιτροπή συμπεριλαμβάνει ε, υποθέσει που καταγγέλει οποιοδήποτε άτομο, η ομάδα περσόνα ή οσδήποτε ΜΚΟ που είναι αναγνωρισμένοι νομικά σε ένα ή περισσότερα από 35 κράτη-μέλη τη οργάνωση. Μόνο τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη τη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απολαμβάνουν το δικαίωμα να υποβάλουν υποθέσει στο δικαστήριο και το δικαστήριο έχει μόνο δικαιοδοσία να εξετάσει υπόθεση από τη στιγμή που η Επιτροπή έχει εξαντλήσει την ιονή δικαστική τη δραστηριότητα. Γι' αυτό πρόσβαση στο δικαστήριο εξαρτάται από την απόφαση τη Επιτροπή όσον αφορά το παραδεκτόν ή όχι τη υποθέσεω και τι αποφάσεω αυτού κατά πόσο υπάρχουν λόγοι για προσφυγή στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Το δικαστήριο ε, έχει συμβουλευτικέ ε, δικαιοδοσίε και την επίλυση διαφορών. Όσον αφορά συμβουλευτική ε, δικαιοδοσία σε περίπτωση διαφορών, ε, ερευνά κατά πόσο έχουν συμμορφωθεί τα κράτη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και δίνει συμβουλές. Οπότε ανταποκρίνεται στι έρευνε που έκαναν φορεί οργαν, του οργανισμού ή των κατών μελών ω βάση συμβατότητα τη εσωτερική νομοθεσία με την Αμερική Σύμβαση ή την ερμηνεία τη συμβάσεως ή άλλων διαμερικανικών εργαλείων. Σύμφωνα, ε, το δικαστήριο έχει δώσει 24 συμβουλευτικέ γνωμοδοτήσει για διάφορα νομική φύσεως θέματα. Το, τα διαμερικανικά εργαλεία και ερμηνεία τη Επιτροπή και το δικαστήριο αυτών έχουν δημιουργήσει πρότυπο όσον αφορά τι υποχρέσει των ανθρώπινων δικαιώματων από τα κράτη και τα όρια που αποφασίζουν οι φορεί, βάσει των ορίων που έχουν αποφασίσει. Παρόλο που οι, οι πρακτικέ ε, δημιουργούν και του νόμου, το Διαμερικανικό Δικαστήριο ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προωθήθηκε από διάφορε αποφάσεις και προωθήθηκε, δόθηκε πιο εξελιγμένη ερμηνεία τη νομοθεσία η Επιτροπή και το Δικαστήριο έχουν θετήσει ερμηνείες όσον αφορά τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται εντός των ιδρυτικών εργαλείων. Σχετικά με αυτό το Δικαστήριο έχει γράψει ότι η ερμηνεία πρέπει να θεωρήσει ότι ε, τις αλλαγές που έχουν γίνει με την πάω του χρόνου και ποιες είναι οι παρούσες συνθήκες. Επίσης, έχει παρατηρήσει ότι η ερμηνεία άλλων διεθνών προδιαγραφών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιοριστεί η απόλαυση και η άσκηση ενός δικαιώματος και θα πρέπει η ερμηνεία να συμβάλλει στην πλέον θετική και ευνοϊκή εφαρμογή μέσω της ερμηνείας. Κατά διάρκεια των 90 χρόνων, ε, τα κράτη της Αμερικής έχουν ένα σταθερό σύστημα προστασίας και πρόθεσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, μέσω της εντολής αυτής, το Δικαστήριο και η Επιτροπή είχαν σαν σημείο αναφορά στην καθολική διακήρυξη, τα σύμφωνα ε, και τους κανόνες που ανέπτυξαν οι διάφοροι φορείς και τι διάφορε διαδικασίε ε, που ήταν πηγή των αποφάσεων. Πιο μόνιμη συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπή και του συστήματο του ΟΗΕ δημιουργήθηκε μέσω της εγκρίσεω κοινή διακήρυξη μεταξύ τη ε, ΕΠΑ, τη Αρμοστία για Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και τη Διαμερικανική Επιτροπή, και αυτό έγινε το 19, του 2014. Στο πνεύμα τη αλληλεγγύη, η Διαμερικανική Επιτροπή επίση δημιουργήσει μηχανισμό συνεργασία με την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ώστε να προωθηθεί η ανταλλαγή των εμπειριών και να υπάρξουν κοινέ δραστηριότητε. Σήμερα η Διαμερικανική αυτή επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει την ισχύ και αξία τη καθολική αντιδιακήρυξη. Όπω αναφέρεται στο προήμιο και τη χάρτα του ΟΗΕ τη Καθολική Διακήρυξη, τα Αμερικανικά κράτη έχουν επανεπεβεβαιώσει την πίστη του στα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπινα, στην αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου και τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών που και προσπαθούν να προωθήσουν την κοινωνική πρόοδο και κανείτε πρότυπα για τη ζωή και οι μεγαλύτερε ελευθερίε. Ευχαριστώ. Thank you, Professor Garcia, Ευχαριστώ πολύ. Από την Αμερικανική Ήπειρο περνάμε στην Αφρική ο καθηγητής κ. Λούμπο. Bonsoir à tous. Ευχαριστώ τους οργανητές του διαλόγου αυτού πολύ καλού επίπεδου και στην οποία έχει προσκληθεί και η Επιτροπή την οποία έχω την τιμή να εκφράζω ε, σήμερα εδώ, να εκπροσωπώ σήμερα εδώ ως Επίτροπος ε, και υπεύθυνο για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Ταγιάννη και τον κύριο Σταύρο Λαμπρινίδη. Επαναλαμβάνω ότι ο Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας, η Αφρικανική Ένωση μάλλον, έχει γιορτάσει και αυτή τα 70 χρόνια από την διακήρυξη και σε επίπεδο του Φόρουμ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ε, και στα πλαίσια της επίσημης συνεδρίασης της Ολομέλειας της Επιτροπής μας. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που στο παρελθόν είχαν δουλέψει πολύ για την συγκεκριμένη διακήρυξη και να ευχαριστήσω επίσης κάποιες προσωπικότητες που χαρακτήρισαν την εποχή τους όπως ο Ρενέ Κασάν για τη Γαλλία, ο Πι Τσάνγκ για την Κίνα, ο Φερνάντε Ούς για το Βέλγιο, ο Σάντα Κρούς για τη Χιλή, ο Τσάρλς Μαλίκ για το Λίβανο, η κυρία Ντελάινο Ρούσβελτ για τις Ηνωμένε Πολιτείες και ο Τζον Χάμπρι για τον Καναδά. Όπως και για όλα τέτοια συμβάντα, οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια της διακήρυξης για τα δικαιώματα μας δίνει την ευκαιρία να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι επιτυχίες, ποια είναι τα λάθη και οι αποτυχίες και να δούμε ποιο είναι το μέλλον ε, για την διεθνή προστασία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα πρέπει να επαναλάβουμε φυσικά την προς την ε, πίστη μας τις αρχές οι οποίες ε, ε, ενέπνευσαν τη διακήρυξη αυτή. Ήταν περιορισμένη η συμμετοχή της Αφρικής βέβαια σε εκείνη την εποχή αλλά εκείνη την εποχή μόνο τρεις αφρικανικές χώρες πήραν μέρος στις προπαρασκευαστικές εργαστίες που έγινε για του κειμένου του 1948. Η Λιβερία ήταν υπέρ, όπως και άλλες 48 χώρες. Η Νοτιοαφρικανική Ένωση τήρησε στάση αποχής και η Αίγυπτος είχε εκφράσει επιφυλάξεις για φιλοσοφικούς λόγους. Πρέπει να θυμίσουμε ότι καμία χώρα δεν τα είχε καταψηφίσει και εμείς στην Αφρική θεωρούμε ότι η δήλωση αυτή, η διακήρυξη αυτή ήταν η πρώτη έκφραση των δικαιωμάτων και των των ελευθεριών των μελών της ανθρωπότητας. Ε, επηρέασε την ανθρωπότητα σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα και προσπαθήσαμε έτσι να προωθήσουμε τις ιδέες αυτές σε όλους τους λαούς και σε όλα τα έθνη έτσι ώστε να οργανωθεί και να αναγνωριστεί η σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη δημιουργία του Οργανισμού Αφρικανικής Ένωσης το 1965 και δηλαδή 17 χρόνια αργότερα τα αφρικανικά κράτη επιβεβαίωσαν την πίστη τους στην διακήρυξη αυτή λέγοντας ότι είναι μια καλή βάση για την ειρηνική συνεργασία και ε, ευνοεί την διεθνή συνεργασία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Αφρικανική Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1981 θεωρείται όπως η, σαν η έκφραση της βούλησης των κρατών ε, μελών της Αφρικανικής Ένωσης ε, να συνεισφέρουν στην καθολικότητα του χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τέσσερα βασικά απαιδεία... Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο για να τα αναλύσουμε. Καταρχάς η δήλωση αυτή, η διακήρυξη αυτή ήταν βασική πηγή έμπνευση ε, για τους συντάκτες της Αφρικανικής Χάρτας. Η Αφρικανική Χάρτα ενίσχυσε πιστεύουμε το περιεχόμενο ορισμένων προβλέψεων της ε, <clears throat> διακήρυξης αυτής. Τρίτον, υπάρχει μια πλούσια και πολύμορφη συνεργασία ανάμεσα στους αφρικανικούς μηχανισμούς ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους αντίστοιχους των Ηνωμένων Εθνών. Και τέλος η, βασική, ε, η τέταρτη βασική ιδέα είναι ότι η διακήρυξη ακόμα και εκεί που δεν είχαν γίνει δεκτές οι προτάσεις δημιούργησε τις δυνατότητες ε, του διαλόγου που υπάρχει σήμερα σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι μία από τις εντολές τις οποίες έχει σήμερα η Αφρικανική Επιτροπή. Είναι η βασική θα έλεγα χάρτα έμπνευσης ε, της Αφρικανικής Χάρτας. Είναι η μήτρα από την οποία βγήκε η Αφρικανική Χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρώτη πηγή έμπνευσης η διακήρυξη όπως ακριβώς και η Αφρικανική Χάρτα είναι ένα συμβιβαστικό κείμενο ε, πάνω στο περιεχόμενο του οποίου συναντώνται διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες και θα υπογραμμίσουμε εδώ ότι το περιεχόμενο των προβλέψεων της διακήρυξης είναι πιο περίπλοκο και πιο ακριβές από τα άρθρα της Αφρικανικής Χάρτας που είναι κάπως γενικόλογοι αλλά συνοδεύεται και από περιοριστικές ρήτρε. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η Αφρικανική Χάρτα έγινε αντικείμενο επεξεργασίας κάτω από πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούσαν μονοκομματικά ουσιαστικά καθεστώτα. Ένας μεγάλος αριθμός των προβλέψεων της Αφρικανικής Χάρτας στην ουσία είναι μια εκ νέου εγγραφή ή προσαρμογή των αντίστοιχων άρθρων της διακήρυξης το άρθρο 2 σαν παράδειγμα της Αφρικανικής Χάρτας στην ουσία επαναλαμβάνει το πρώτο τμήμα της παραγράφου 1 της δήλωσης, της διακήρυξης. Ε, θα δείτε ότι στην ουσία έχουμε γράψει με διαφορετικό τρόπο αυτό που λέει η διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ίδιο θα γίνει και για τα υπόλοιπα άρθρα. Θα δείτε ότι στην ουσία πρόκειται για κάποιες προσαρμογές ή εκ νέου καταγραφές. Ε, δεύτερον θα ήθελα να πω ότι στην ουσία ε, ε, εννέα από τους συντάκτες, ε, ε μάλλον κάποιος από τους συντάκτες, ο Ρενέ Κασά, είχε πει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τρίπτυχο. Το κεντρικό είναι η διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι άλλες δύο πτυχές ήταν οι επιμέρους συνθήκες και τα εφαρμοστικά μέτρα. Το ίδιο ακριβώς μπορούμε να πούμε ε, και για την Αφρικανική Χάρτα, ότι είναι κάτι το οποίο βοηθά τον καθολικό χαρακτήρα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η τρίτη βασική ιδέα είναι η σωστή και πολύμορφη συνεργασία ανάμεσα στον ε, Οργανισμό τον Αφρικανικό και τον Ηνωμένα Έθνη Καταρχάς ο βασικός λόγος είναι ότι τα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει τη συμφωνία αυτή έχουν αναλάβει να σεβαστούν ακριβώς τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Και τέλος έχουν ανοίξει και νέα πεδία στον τομέα του περιβάλλοντος, της γενετικής κληρονομίας Νομίζω ότι μπορούν όλα αυτά να διερευνηθούν και μέσω των περιφερειακών και των, των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Ας πούμε τι γίνεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, με την χρήση ε, μη επανδρομένων ε, εναερίων μέσων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας τι γίνεται σε σχέση με την, τον σεβασμό της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Και η τελευταία ιδέα είναι ότι η διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι κάτι το οποίο εμπνέει ε, τις αντίστοιχες αφρικανικές ρυθμίσεις. Το, το άρθρο 47 της Αφρικανικής Χάρτας δίνει στον οργανισμό και στην Επιτροπή την αποστολή της διασφάλισης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό περιλαμβάνεται ουσιαστικά και στην αρχική διακήρυξη. Η συζήτηση για τα δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνονται στην διακήρυξη ε, οδηγεί σε τρία συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι στην αρχική πρόταση ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπήρχε ένα άρθρο 20 το οποίο έθετε την αρχή της αναφοράς και επικοινωνίας. Το χρησιμοποιούμε αυτό στην Αφρική. Δεύτερον, υπήρχε ε, και ε, το άρθρο 38 που δεν είχε γίνει δεκτό και είχε προτείνει ο Ενεκασά που πρότεινε ένα σύστημα προσφυγής και έφεσης διοικητικό ή δικαστικό και αυτό το χρησιμοποιούμε στην Αφρική. Και τέλος, δεν έχω πια πολύ χρόνο, ε, υπήρχε επίσης ε, στο ε, τμήμα που απορρίφθηκε μια άλλη πρόβλεψη την οποία, η οποία ζητούσε οι χώρες ε, να λάβουν επιπλέον μέτρα και διεθνείς συμβάσεις για τον σεβασμό α, της συγκεκριμένης Εδώ μπορούμε να πούμε ότι δεν είχαν γίνει δεκτές οι προτάσεις αυτές, αλλά μας έχουν βοηθήσει να κάνουμε αυτό για το οποίο είμαστε εδώ σήμερα και σε επίπεδο αφρικανικό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Thank you, Professor Ευχαριστώ καθηγητά Λούμπου για την ε, αφρικανική αυτή οπτική γωνία. Καταζήνα καταπλάτσε, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το δικό μας γραφείο είναι ιδιαίτερα περήφανο που βρίσκεται εδώ και εκπροσωπείται από εμένα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σας μιλήσω όμως για αυτό το γραφείο των, δικαιωμάτων των δημοκρατικών θεσμών, αλλά θα ήθελα να εστιάσω σε ένα από τα ερωτήματα για το πάνελ, δηλαδή πώς θα έρθουμε σε επαφή με ευρύτερα στρώματα τη κοινωνία και θα του πούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι. Υπάρχουν κάποιε αντιλήψεις ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να του δώσουμε μεγάλη προσοχή. Αυτά τα λέω όχι μόνο γιατί είμαι ψυχολόγος, αλλά γιατί πιστεύω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς. Θέλουμε ε, να πιστεύουμε ότι το σημαντικό είναι αυτό που λέμε στον κόσμο για τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα είναι όμως τι ακούνε και τι καταλαβαίνουν οι συνανθρωποί μας. Αυτό για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως. Να δώσουμε ανθρώπινο πρόσωπο στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Στη δέκατη επέτειο της ε, ε, διακήρυξης ε, είπε κάποια πράγματα η Έλληνα Ρούσβολτ, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Είπε όμως μεταξύ άλλων ότι τα οικομενικά ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα έχουν νόημα πουθενά αν δεν έχουν νόημα για τον κάθε άνθρωπο στον ιδιωτικό του κόσμο και πολλά το επιβεβαιώνουν έρευνες από το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα. Σε μια έρευνα μελετήθηκε η αντίληψη των ανθρώπινων δικαιώματων και μια ομάδα του 40% περίπου που είχαν κάποιε αντικρουόμενε στάσει και συμπεριφορέ δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώ τα οικομενικά ανθρώπινα δικαιώματα είχαν την οποιαδήποτε σχέση με την καθημερινότητά του. Όταν έγινε όμω αυτή η διασύνδεση, έγιναν υποστηρικτέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε μια άλλη έρευνα ή πολλέ ε, στην πολιτική ψυχολογία που λένε ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους ως άτομα. όσο μεγαλύτερο είναι ο αριθμό δεν θα υπάρξει συνέστηση όταν από το να πάμε στους δύο. Σάκι κνάμπινγκ λέγεται αυτό στα, στην αργό ε, των ε, ψυχολόγων. Αμβλύνεται δηλαδή εν συνέστηση όσο μεγαλύτερη είναι η αριθμή. Γιατί διεθνεί συμβάσει, γιατί τα διεθνομικά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικά, τι σημαίνουν τελικά για τον καθένα μα, Πώ μπορούμε αυτά να τα συσχετίσουμε με την καθημερινότητα και τα προσφυλή ζητήματα για όλους μας. Σίγουρα πρέπει να σταματήσουμε την αφηρημένη ε, ορολογία και θα σας δώσω ένα παράδειγμα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 καταλάβατε οι γυναίκες να έχουν περισσότερες δυνατότητες και να είναι πιο ίσες πλέον. Σας συγχαίρω να το πιάσατε από αυτό που σας διάβασα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να μην χρησιμοποιούμε ε, αριθμούς, εκατομμύρια που εκτίθενται στο ρατσισμό κτλ. Δεν πρόκειται να νιώσει συνέστηση ο συνανθρωπός μας με αυτά. Επίσης υπάρχει υπερβολική εξειδίκευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ε, λέγεται. Όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, ο μόνος παράγοντας ε, που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη είναι η ανθρώπινη φύση. Γιατί η κομμουνικότητα σημαίνει όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ε, δικαιώματα. Και αυτά πρέπει να εφαρμόζονται. Δικαιώματα των γυναικών, των μειονοτήτων, των μεταναστών, ε, τα αντιμετωπίζουμε σαν να είναι διαφορετικά από αυτούς που δεν είναι μετανάστες γυναίκες ή ε, μειονότητες. Φυσικά πρέπει να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τις ευάλωτες ομάδες και γι' αυτό απαιτείται συνεχής προσπάθεια. Όμως όταν ειδικεύουμε, εξειδικεύουμε το μήνυμα και μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα συγκεκριμένων κατηγοριών, δημιουργούμε την αντίληψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ανήκουν μόνο σε κάποιου. Και επομένω, γιατί μα εκπλήσει όταν έρχονται κάποιοι και μα λένε το μόνο που σα νοιάζει είναι οι μετανάστες και οι Ρωμά και για μας δεν δίνεται δεκάρα. Ούτε να εξειδικεύουμε το δικαίωμα. Σε σχέση δηλαδή με την αστική πολιτική συμμετοχή, τη θρησκευτική ελευθερία κτλ. Δεν είναι καλό να τα αφήνουμε εκτό του οικουμενικού πλαισίου γιατί δημιουργούμε το δικαίωμα ότι είναι κάποτε διαφορετικό αυτό το δικαίωμα από κάποια άλλα. Και άρα ότι μπορεί να είναι επιλεκτικά, να υπάρχει ε, ε, επιλεκτική χρήση και σεβασμό των δικαιωμάτων. ανθρώπινα δικαιώματα πολλές φορές παρουσιάζονται ως εμπόδιο στο να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα της πλειοψηφίας απέναντι στη στάση κάποιων μειοψηφιών. Άρα κάποιοι πιο σημαντικοί από κάποιους άλλους. Υπάρχει επιλεκτική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή τα δικαιώματα κάποιων μπορεί να είναι ε, σεβαστά σε βάρος άλλων. Ή η μεροληψία αρνητικής παρουσίασης. Ακούσαμε κάποιες προσωπικές ιστορίες. Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες. Gapminder είναι ένα project ε, του γιατρού Ρόσλινγκ. Έχετε δει ίσως ότι στον Ταβός ε, αναφέρονται μόνο αρνητικά και δεν ε, βλέπουν κάτι θετικό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης μεροληψίας αυτής. Μεροληψίας του πιστεύω, της ε, έλλειψης αναλυτικών δεξιοτήτων ή από τα μέσα ενημέρωσης που δίνουν μεγάλη σημασία στα ασυνήθιστα. Αν δείξουμε στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άποψη κάποιου, η άποψη αυτή ενισχύεται. Το ίδιο θα συμβεί όμως αν δώσουμε τα αντίθετα επιχειρήματα. Μεροληψία της επιβεβαίωσης λέγεται αυτό. Αν θέλουμε να καταρρύψουμε ένα μύθο, κάποιος θα κολλήσει εκεί και όχι στο επιχείρημα που τον καταρρύπτει παραδείγματο χάρη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και με πολλά μηνύματα που περνάμε ενισχύεται αυτή η αρνητική ημεροληψία. Ούτε θα αλλάξει συμπεριφορά με βάση τα δεδομένα και τις στατιστικές. Και αυτό είναι ένα που κάνουμε πολλές φορές. Γιατί είναι πολύπλοκοι παράγοντε που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ένα από του σημαντικού παράγοντε που καθορίζουν τι ανθρώπινε αξίε, την ανθρώπινη συμπεριφορά, ε, είναι παραδείγματος χάρη φορές και τα σύμβολα. Και το δείχνουν αυτό πολλές μελέτες. Στους περιφερειακούς ή διεθνείς οργανισμούς πολλές φορές η γνωστική ψυχολογία παραγνωρίζεται εντελώ. Και το επίκεντρο είναι πιο πολύ τα αρνητικά. Δηλαδή μιλάμε για παραβιάστροπη δικαιωμάτων, προκλήσεις σε ό,τι αφορά την προστασία τους. Φυσικά και αυτά είναι πραγματικά φαινόμενα και πρέπει να τα πούμε και να τα βροντοφωνάξουμε. Δεν θα πρέπει όμως το ίδιο να κάνουμε με θετικά παραδείγματα προόδου, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο Πίτσμπεργκ, ε, στις πυροβολισμού που έπεσαν εκεί, όλοι καταδίκασαν ε, την αποτρόπαια πράξη. Δύο μέρες μετά η μουσουλμανική κοινότητα του Πίτσμπεργκ συγκέντρωσε πάνω από 100.000 δολάρια Αμερικής για να στηρίξει τα ε, θύματα, ε, τους Εβραίους που χάθηκαν. Αυτό θα πει αλληλεγγύη, θα πει ε, μέρημνα. Αυτά τα λέει και η Οικομενική Διακήρυξη. Τα ακούσαμε το ίδιο. Πολύ ε, βρωτοφωνάξαμε την υποστήριξή μας αυτή την πράξη αλληλεγγύης. Όταν επιλέγουμε λοιπόν αρνητική γλώσσα κυρίως, όταν μιλάμε για τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς να το θέλουμε δημιουργούμε μία αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι σημαίνουν προβλήματα. Αντί δηλαδή να ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για ασφάλεια, για ελπίδα, ενισχύουμε το φόβο του κόσμου. Όποιος νιώθει φόβο ανασφάλεια θα πέσει εύκολα θύμα των λαϊκιστών που χαϊδεύουν τα αυτιά τους. Είμαστε ε, σε μια επικίνδυνη εποχή κόποση ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν εστιάζουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα ω ε, ε, πρόβλημα, θα είμαστε σαν το Βοσκό που έλεγε ότι έρχεται λύκο να το φάει τα πρόβατα και τελικά δεν το πίστευε κανένα όταν αυτό ήταν αλήθεια. Και φυσικά αυτό θα οδηγήσει σε κινησμό και αδράνεια. Τέλος. Είμαστε σε ένα echo chamber Δηλαδή ε, δημιουργείται απήχηση, αντίχηση μάλλον, ε, αντίλαλος σε αυτό το χώρο που είμαστε. Πρέπει λοιπόν να βγει προς τα έξω αυτό. Να μην μιλάμε μόνο με τους ίδιους ε, εμπειρογνώμενους, καθημερινούς φορείς ε, κτλ. Η ΟΑΣΕ λέγεται από πολλούς ως γραφείο σεμιναρίων. Μπορεί να είναι αστείο για κάποιους αυτό, αλλά πρέπει να είναι καμπανάκι για μας και να μας ξυπνήσει. Πρέπει να βγούμε προς τα έξω, να γίνουμε, ε, να μας ακούσουν και οι άλλοι που δεν μας ακούν ακόμη. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κοινό χώρο. Υπήρχε σε μια μελέτη αρχιτεκτονική του πώς να μιλά κανείς. Architectural speaking. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί όλα τα σωστά εργαλεία. Όμως 80% των ε, μέσων που χρησιμοποιούν οργανώσεις για τη δημόσια επικοινωνία πάνε στη διανομή των πληροφοριών από την κορυφή προς τη βάση για την οργάνωση. Και κλείνω με μια πρόταση. Τι θα συμβεί αν του χρόνου το 19 αντί να οργανώσουμε άλλη μια διάσκεψη, άλλο ένα σεμινάριο οι περιφερειακοί μηχανισμοί, οι διεθνείς οργανισμοί βάλουν τα κονδύλια σε ένα κοινό κορβανά, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε πιο αποτελεσματικά ε, και να είναι οικομενικά κατανοητά τα μηνύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καραπχάτσεφ. Πολύ σαφή αυτά που είπατε. Μπράτο Ρούντολφ, έχετε το λόγο, συμπατριώτη μου τη Γερμανία. Εξοχότητε συγκεκριμένα μέλη, είναι χαρά για μένα που είμαι εδώ σήμερα μαζί σα για την ευδικοστή επέτειο των οικουμενικών δικαιωμάτων. Είδαμε μεγάλη πρόοδο από όταν υιοθετήθηκε το 1948. Επίσης βλέπουμε να υπάρχει μια επίθεση κατά ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πλαισίου Διεθνού Προστασία. Θα προσπαθήσω τώρα να δείξω πώ οι εθνικοί θεσμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα είναι ράιλ, υποστηρίζουν την καθολικό χαρακτήρα και την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξασφαλίζοντα ότι θα το λαμβάνουν υπόψη, θα στερνιστούν οι ντόπιοι τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και θα μπορούν να ενταχθούν ε, μαζί με τι ε, αξίε Ευρωπαϊκή Ενώσεω. 70 χρόνια πριν, μετά από δύο καταστροφικούς παγκοσμίους πολέμους, η εθνική κοινότητα αναγνώρισε στην Οικουμενική Διακήρυξη ότι η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη και η ανάπτυξη θα ήταν εφικτά μόνο μέσω του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία είναι καθολικά από τη φύση του, οικουμενικά και ε, δεν είναι αναγνωρισμένα για, εκείνους για όλους. Λοιπόν, αυτό το κοινό πρότυπο των επιτευμάτων τελικά έγινε ε, καθολική αξία. Πριν από 25 χρόνια, η Παγκόσμια Διάσκεψη τη Βιέννη για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναγνώρισε ότι οι περισσότερε προσπάθειε έπρεπε να καταβληθούν, τόσο ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα να γίνουν μια επιτόπια πραγματικότητα. Για αυτόν τον σκοπό, οι χώρε δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την εσωτερική εφαρμογή και το σχετικό μηχανισμό και το μηχανισμό λογοδοσίας και κυρίως κάλεσαν κάθε κράτος να δημιουργήσει ένα φορέα που θα υποπτεύει και θα συμβουλεύει όσον αφορά την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και να προωθεί έναν πολιτισμό, μια κουλτούρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο εποπτικός μηχανισμός ε, παρα, παρακολουθούσε την κατάσταση στη χώρα και έπρεπε να λογοδοτεί στο γενικό κοινό και το κοινοβούλιο να ερευνά τις καταστάσεις για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και τελικά να προσφέρει στα δικαστήρια τα διεθνή και τα τοπικά για παραβιάσεις ε, και να εξετάζει καταγγελίες αρμόδιες φορές των Φιλιππίνων ερευνά εξοδικαστικές δολοφονίες συλλέγοντας στοιχεία για μελλοντικέ ε, ποινικέ ε, διαδικασίες δικαστικές. Οπότε υπάρχει ο κατάς μηχανισμός για να παρεμποδίζονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διεθνώς πρότυπο ε, είναι οι αρχές του Παρισίου που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ πριν από 25 χρόνια. Σήμερα η ύπαρξη των αρχών ε, των Παρισίων και φορέα που συμμορφώνεται με αυτό είναι ε, μέσα στον στόχο 16 της ε, θεματολογίου για βιώσιμη ανάπτυξη του 2030. Είναι ανεξάρτητοι φορεί αυτοί από την κυβέρνηση με μια εντολή να προωθούν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, διαπιστεύονται κάθε πέντε χρόνια με αναφορά στι αρχέ των Παρισίων για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία του, ο πλουραλισμό, η λογοδοσία και η αποτελεσματικότητα. Σήμερα υπάρχει η Παγκόσμια Συμμαχία των Εθνικών Θεσμών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που αποτελείται από τέσσερα περιφερειακά δίκτυα Αφρικής, Αμερικανικής Υπήρου, Ασίας, Ειρηνικού και Ευρώπης. Αυτοί οι εθνικοί φορεί για ανθρώπινα δικαιώματα γεφυρώνουν το διεθνέ επίπεδο με το, με το εσωτερικό. Εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ουσιαστικά είναι εθνικοί φορεί που κατανοούν ποια είναι η τοπική ιδιαιτερότητα, η εθνική ιδιαιτερότητα με το να βοηθήσουν την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμβάλλουν στην πρόληψη. Πολλοί φορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν συστήματα έγκαιρη προειδοποίηση για καινοτόμα συστήματα μέσω καινοτόμων συστημάτων εποπτεία. Ο αρμόδιο φορέα του Κένια ε, εντόπισε κάποιε ενδεχόμενε περιοχέ για σύγκρουση κατά τη προεκλογική ε, και ε, λάμβανε μέσω SMS πληροφορίε από τον τόπιο πληθυσμό για να μπορεί να αντιδρά γρήγορα. Οι φορεί του ανθρώπινα δικαιώματα επίση αναφέρονται σε διεθνεί φορεί του ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, διευρύνουν και αυξάνουν τον έλεγχο και την ανταπόκριση των φορέων, προωθώντα ταχεία δράση και ε, υποχρεώνοντα λογοδοσία πλευρά κυβερνήσεων. Εν γέννη, αυτοί οι φορεί συμβάλλουν στο έργο περιφερειακών οργανισμών και πλησίων για ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματο χάρη το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τα Εθνικά Ανθρώπινα, ε, το ΕΝΡΙ, ε, που είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Φορετρόπινων Δικαιώματα, έχει μόνιμο καθεστώ μοτίβου παρατηρητού από πρώτου Συμβουλίου τη Ευρώπη, ε, τη Αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου τη Ευρώπη στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στην Αμερικανική ε, Ήπειρο, αυτοί οι φορεί έχουν υποβάλει υποθέσει στη Διεθνή Επιτροπή, την Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρώπινα Δικαιώματα, όταν κινδυνεύουν. Το δίκτυο των Αφρικανικών αυτών φορέων έχει καταρτήσει κατευθείαν γραμμέ για την εποπτεία τη εφαρμογή των συστάσεων τη Αφρικανική Επιτροπή πεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών στην Ειρηνικό και την Ασία ε, ε, λόγω ελλείψης τοπικού πλαισίου ο αρμόδιος φορέας συνεργάζεται εκτεταμένα με την Διακυβερνητική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΑΖΕΑΝ. Αυτή οι φορεί, οι εθνικοί ανθρώπινα δικαιώματα, έχει σημαντικό ρόλο να παίξουν, πλησιάζοντα περισσότερο την κοινωνία για σημαντικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί τη 70η επαιτία, επαιτίο τη ε, καθολική εκεί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια στροφή εναντίον αυτών των δικαιωμάτων. Αυξάνεται ο λαϊκισμό και αυταρχική διακυβέρνηση ε, που καταλήγει σε ένα αφήγημα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο τοπικό και σε επίπεδο ΟΗΕ. Τα κράτη έχουν φύγει από το διαμερικανικό σύστημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συνοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιμετωπίζει προβλήματα και βλέπουμε ότι τελικά αμφισβητείται και εφαρμογή διεθνών προτύπων σχετικά με αυτά τα δικαιώματα. Επίση και η εποπτική λειτουργία των περιφερειακών δικαστηρίων στα ανθρώπινα δικαιώματα αμφισβητείται. Οι τοπικοί φορεί στα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να ελέγξουν αυτέ τι εξελίξει. Αποτελούν από στο στήμα του Διεθνού Συστήματο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρέπει να εφαρμόσουν διεθνή πρότυπα για ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά επίση υπάρχουν και εθνικοί φορεί οι οποίοι ε, πλησιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στου κατόχου των δικαιωμάτων. Έτσι τελικά ενστερνίζονται οι τοπικοί προθεσμοί τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν υποστηρίζουν την εφαρμογή των καθολικών προδιαγραφών σε διάφορα εθνικά πλαίσια και όταν παρέχουν εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον πληθυσμό καθώς και για φορείς του κράτους. Οι εθνικοί φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα φέρνουν στην πατρίδα, στη χώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνεργάζονται στενά με του κρατικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγματι, η δήλωση του Μαρακέ του Γκάνρι και τα περιφερειακά ε, προγράμματα ε, δείχνουν πώς οι φορείς αυτοί μπορούν να προστατεύσουν το δημοκρατικό χώρο στη χώρα και πώς να στηρίξουν τους προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό συμπεραβάνει η πρόληψη και σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε στενή συνεργασία με διεθνείς μηχανισμούς. Το σχέδιο δράση του ΕΝΡΙ ξεκίνησε σήμερα και μπορεί να το βρει κανεί κάτω, στην είσοδο, μαζί με ένα δημοσίευμα που δείχνει το πώ τα NHRI υποστηρίζουν του προσφυστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την ευρύτερη Ευρώπη. Κυρίε και κύριοι, αυτοί ε, οι φορεί οι εθνικοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα ενισχύουν ε, τι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Ενώση να εφαρμόζει αυτά τα δικαιώματα. Εντό των κρατών μελών, οι φορεί αυτέ, με την υποστήριξη του ΕΝΡΙ, κινούνται προ την εφαρμογή τη Χάρτη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Σε τρίτε χώρε, αυτοί οι φορεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα παρέχουν πληροφορίε από επιτόπιο επίπεδο σε αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Ενώση, συμμετέχουν σε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η έκθεση προόδου και διενεργούν και εφαρμόζουν κοινά προγράμματα για να προωθήσουν την ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο συνεργαζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά αυτοί οι φορεί είναι αξιόπιστοι φορεί εντό του μηχανισμού του κράτου και παρέχουν περιθώριο για ανοιχτό διάλογο και ανεξάρτητη δράση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εντό τη εθνική δικαιοδοσία. Ο σημαντικό ρόλο αυτών των εθνικών φορέων έχει αναγνωριστεί στο παρόν σχέδιο δράσεω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία που έχει συνεργασία σαν με τα εθνικά δίκτυα αυτά ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν πρώτη δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει αυτού του φορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω τη συμμορφώσεω με τι αρχέ των Παρισίων συμπεριλαμβανομένων και περιπτώσεων όπου αυτοί οι φορεί εθνικοί απειλούνται, όπω γίνεται αυτό στι Φιλιππίνε ή στη Σιέρα Λεόνε. Πέρα από την πολιτική υποστήριξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τον Γκάνρι και τα περιφερειακά δίκτυα αυτού για να παράσχει δημιουργία δυνατοτήτων και ανταλλαγή με πληροφοριών μεταξύ ομοτήμων συμπεριλαμβανομένων με του ε, φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΝΡΙ. Όμω η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των φορών των εθνικών μπορούσε να ισχυρότερη, του ώστε τα καθολικά δικαιώματα να είναι πραγματικότητα τη πάση. Η συμμετοχή αυτών των εθνικών φορών για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί περισσότερο για βαθύτερη και πιο συνεπή προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικού διαλόγου την περιοδική ε, επιθεώρηση του ΟΗΕ για τα σχετικά θέματα και άλλε διαδικασίε, ούτω ώστε η πρόοδο να μην απολυστεί και αναμένεται ότι το νησιά διαδράσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία συμπεριλάβει του εθνικού φορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο να γνωρίσει αυτού του εθνικού φορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα για βασικού εταίρου να υποστηριχθούν οι αξίε και τα δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω συμπεριλαμβανόντου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δημοκρατικού χώρου. Κυρίε και κύριοι, μέσω συνεργασία αυτή η Εθνική Φορή των Ανθρώπινων Δικαιώματα, η Κοινωνία των Πολιτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξουν το διεθνές και περιφερειακό σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίξει την εθνική εφαρμογή καθολικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικών προτύπων όπως αυτό προβλεπόταν από την καθολική διακήρυξη πριν από 70 χρόνια. Μέσω συνεργατικής δράσης μπορούμε το πολυμερές σύστημα ανθρωπίνων δικαιώματων να το καταστήσουμε πραγματικότητα, να τον ενστερνιστούν τοπικοί πληθυσμοί και να συμμετέχουν σε όλους και να προστατεύουν τους κατόχους των δικαιωμάτων και να έχουμε αποτελεσματικά περιφερειακά δίκτυα. Το Γκάνρι, το Ένρι, και όλα τα εθνικά συστήματα είναι έτοιμα να συνεργαστούν μαζί σας. Και έτσι κάθε άνθρωπος μπορεί να απολαύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα πανταχού. Μέσω καθολικών δικαιωμάτων και αξιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στον τελευταίο για σήμερα ομιλητή καθηγητής Πάλματερ από το Τόροντο. Εκπροσωπώ την περιφέρεια Νίκ Μάγκη, σε αυτό που είναι σήμερα Καναδά. είμαι όμω από τη φυλή των Ινδιάνων Μικ Μάου, από το Ινδιάνικο έθνος Μικ Μάου και ευχαριστώ τον Αντώνιο Ταγιάννη που και τον ε, Αντιπρόεδρο Παντσέρη σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα ως ηθαγενής να μπορέσω να εκφράσω την άποψή μου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλές φορές εμείς μιλάμε για την πρόοδο που έχει γίνει, για τους νόμους και τα λοιπά που είναι ε, βελτιωτικοί και αυτό μας κάνει να είμαστε ικανοποιημένοι, μας κάνει να χαλαρώνουμε ε, και νομίζω ότι δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Είναι μια ανθρώπινη τάση αυτή. Αυτή τη στιγμή κάποιος ε, ακούει κάτι καλό να μένει σε αυτό και να μην βλέπει τα άσχημα. Αλλά παρόλα αυτά οι ηθαγενείς πληθυσμοί επηρεάζονται όχι μόνο από τις κυβερνήσεις, όχι από τις διεθνείς οργανώσεις, Υπάρχει και άλλη μία πλευρά στα μηνύματα τα οποία πρέπει να στείλουμε. Το θέμα είναι να ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε τους ηθαγενείς να έχουν ηγετίδα θέση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δώσουμε ελπίδες στις κοινότητές μας γιατί όταν οι κοινότητές μας δεν έχουν ελπίδες τότε έχουμε πολύ δυστυχώς υψηλά επίπεδα αυτοχειρίας. Πολλές χώρες θεωρούν ότι είναι παραδείγματα για τον υπόλοιπο κόσμο. Όχι μόνο είναι ευχαριστημένες επειδή κάνουν κάποια πράγματα καλά, αλλά περηφανέζονται και στον υπόλοιπο κόσμο γι' αυτό. Θα σας δώσω τον Καναδά σαν παράδειγμα. Είναι μια από τις πιο μεγάλες και πλούσιες χώρες του κόσμου. Σε κάθε διεθνές φόρουμ λέει ότι είναι υπέρ της πολλαπλότητας, του πλωραλισμού, του σεβασμού των φίλων, υπάρχουν ε, επιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις μεγάλες επαρχίες, συμμετέχουμε σε πάρα πολλές ε, μορφές εξουσίας και οργάνωσης, ελευθερία του τύπου και μάλιστα ε, ε, έχει και το δικαίωμα το κράτος της προστασίας της περιουσίας των ηθαγενών. Θεωρείται μία από τις πέντε καλύτερες χώρες για να ζει κανείς και γενικά θεωρείται μία από τις δέκα καλύτερες χώρες στον κόσμο. Είναι απίστευτα καλή η κατάσταση. Όταν όμως απομονώνεται τις συνθήκες ζωής των ηθαγενών στον Καναδά τότε βλέπεις, βλέπετε ότι ο δίκτυς ανάπτυξης από τις πρώτες 10 θέσεις πηγαίνει στην 60η θέση μαζί με χώρες όπως ε, Αργεντινή και τα λοιπά. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια τρομακτική εσωτερική αντίφαση στη χώρα μας. Ο προηγούμενος ε, εισηγητής του τους λέει ότι ο Καναδάς συνιστά μια τρομακτική αντίφαση ουσιαστικά. Είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρητικά προστατεύει με νόμους τους ηθαγενείς και όμως έχει διαπράξει παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα προστασίας. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας τομέας προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που να μην παραβιάζεται από τον Καναδά σε σχέση με τους ηθαγενείς. Μερικές φορές λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και να αναφερόμαστε σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Οι ηθαγενείς είναι το 5% του πληθυσμού ε, στον Καναδά, αλλά το 20% από αυτούς δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό σε μια τόσο πλούσια χώρα το 40% των αστέγων στον Καναδά είναι ηθαγενείς και όταν δείτε σε συγκεκριμένες επαρχίες φτάνει και το 90%. Έχουμε πραγματικά ε, μαζικά επίπεδα ανεργίας εδώ και δεκαετίες. Είχαμε επίσης ε, εξαιρετικά ασχήμα επίπεδα υγείας ε, και ο πρώτος λόγος αιτία θανάτου, η πρώτη για τους νέους μας είναι οι αυτοκτονίες. Οι ηθαγενείς του Καναδά και το επιβεβαιώνω αυτό εδώ και 35 χρόνια έχει το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών. Πώς μπορεί κανείς να το αγνοήσει κανείς αυτό, για τις γυναίκες και τα παιδιά τα πράγματα είναι χειρότερα. Το 60% των οικογενειών των ηθαγενών ζουν σε πλήρη έμβια. οι η υπερβολική παρουσία θα έλεγα των ηθαγενών στις φυλακές δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει σε όλες τις ηλικίε, σε ορισμένα σοφρονιστικά ιδρύματα το 98% είναι Ινδιάνοι, είναι ηθαγενείς και έτσι λοιπόν ο Καναδάς λέγεται δείχνει προς τα έξω ότι προχωρά και προοδεύει αλλά αυτό δεν ισχύει ε, για τους ηθαγενείς. Επίσης ε, τα ποσοστά των δολοφονιών γυναικών και των ε, γυναικών που αγνοούνται είναι τεράστια τα ποσοστά αυτά και είναι κάτι το οποίο δεν θα συνέδεε κανείς στον Καναδά. Το 40% των γυναικών, κορίτσια, γυναίκες, παιδιά πέφτουν θύματα απαγωγής για έναν και μόνο λόγο ε, γιατί δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχουν συνέπειες στις κοινωνίες μας για τη βία εις βάρος των γυναικών ηθαγενών. Υπάρχουν ε, οργανώσεις όπως το Human Rights Watch, η Amnesty International μας βοηθούν, προσπαθούν να φέρουν όλα αυτά στην προσοχή του υπόλοιπου κόσμου. Και αν δεν είχαμε τους διεθνείς μηχανισμούς τότε πραγματικά οι φωνές μας δεν θα πήγαιναν πουθενά. Για πάρα πολλά χρόνια προσπαθήσαμε να ζητήσουμε από τον Καναδά να αναλάβει δράση. Αλλά παρόλα αυτά οι διάφορες επιτροπές οι οποίες δημιουργήθηκαν, οι επιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σώματα τα οποία μας έδωσαν την δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να κάνουμε ορισμένες συστάσεις και για να ενθαρρύνουμε τελικά τον Καναδά να αλλάξει τα πράγματα. Γι' αυτό νομίζω ότι οι παγκόσμιοι μηχανισμοί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο απαιτείται. Έχουμε να κάνουμε με μια ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει φυσικά στην ιστορία βλέπουμε κάποιες απεικιοκρατικές αντιλήψεις αλλά έχουμε περάσει από πάρα πολλά δυστυχώς ε, στηρώσεις υποχρεωτικές ε, δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα τέτοια φαινόμενα σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις στη χώρα μου ενώ δεν υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσμο πια υπάρχουν πολλοί οι οποίοι φυσικά ασκούν κριτική και στα Ηνωμένα Έθνη και στους άλλους μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα διότι δεν έχουν ε, μηχανισμούς επιβολής, δεν έρχονται με το στρατό τους σε βάση περιπτώσει έτσι ώστε να εφαρμόσουν αυτά τα οποία πρεσβεύουν. Αλλά αν δείτε τι γινόταν το 1970 όταν ο Καναδάς είχε αρνηθεί να ανακαλέσει νόμους οι οποίοι δεν σεβόντουσαν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό είναι φυσικά μία παραβίαση της, της, του, του σεβασμού των, των ίδιων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των σεβασμών. Και κανένα διεθνές σώμα δεν εξέτασε αυτό και δεν, κανένας διεθνής οργανισμός δεν βγήκε να πει ότι δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά στις γυναίκες των Ιθαγενών. Επίσης οι εθνικές έρευνες οι οποίες γίνονται για τις γυναίκες που χάνονται, που χάνουν τη ζωή τους. Υπήρξαν, υπήρξαν μορφές αλληλεγγύης από ηθαγενείς στις Ηνωμένε Πολιτείε, από Ινδιάνους δηλαδή, από τις Ηνωμένε Πολιτείε ή από το Μεξικό που μας βοήθηκαν και πράγματι διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια σοβαρότατη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στον Καναδά και θα έπρεπε να ξεκινήσει μια έρευνα. Α, υπήρξαν όμως τεράστιες αναβολές, υπήρξε τρομακτική καθυστέρηση και χρειάστηκε τρομερή πίεση για να ξεκινήσει επιτέλους ε, μια έρευνα η οποία συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δεν θα το είχαμε πετύχει αυτό αν δεν υπήρχαν οι διεθνείς μηχανισμοί οι οποίοι μας βοήθησαν να ακουστούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση προς όλους εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βλέπουν το τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες. Να μην μένουν σε αυτά που λένε οι ειδήσει, αλλά κυρίως σε αυτά που δεν λένε οι ειδήσει. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Καναδά θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν σας ενδιαφέρουν. Όχι, έχουμε να κάνουμε με μια παγκόσμια οικογένεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικού χαρακτήρα και φυσικά ε, ε, εμείς είμαστε με τον τρόπο μας υπεύθυνοι για τις εξελίξεις στον κλάδο αυτό και εμείς από τις χώρες μας θα πρέπει να ζητήσουμε από τις υπόλοιπες χώρες να σέβονται τις ε, διεθνείς ρυθμίσεις. Όταν υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ινδιάνων στον ε, ε, Καναδά σαν παράδειγμα για να εξυπηρετηθούν εμπορικοί στόχοι ή στόχοι που ορίζονται από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες είναι κάτι το οποίο αφορά και σε άλλες κοινότητες ε, ηθαγενών σε άλλες χώρες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Καναδάς ή κάθε χώρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η ανθρωπότητα μοιάζεται για όλα αυτά γιατί πρόκειται για παγκόσμια ε, συλλογικά φαινόμενα. Το θέμα δεν είναι τι τίτλο έχει σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει σημασία το τι επίπεδα θεωρητικά προστασίας έχει κανείς. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις αυτές και πώς επηρεάζουν άμεσα τους λαούς οι οποίοι βιώνουν τις συνέπειες αυτών των πολιτικών. Συνεπώς λοιπόν δεν θα πρέπει να πιστεύετε ότι είναι ένα αγώνας δημοφιλίας τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου ο καθένας προσπαθεί να γίνει πιο αρεστός βελτιώνοντας τυπικά τον σεβασμό τους. Thank you, Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ συγκινητικά αυτά που μας είπατε. Θα γνωρίζετε ίσως ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωκοινοβουλίου επισκέφθηκε τον Καναδά. Πριν από δύο εβδομάδες μάλιστα. Και διάβαζα τις πρώτες ε, αναφορές προσφάτως. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει το αργότερο 7 και 5, 7 και 10 να έχουμε ολοκληρώσει. Άρα έχουμε γύρω στα 25 λεπτά. Requests to speak. Παρακαλώ, όσοι έχετε ζητήσει το λόγο, να είστε σύντομοι δύο λεπτά, ώστε να μπορέσουν ε, και τα μέλη πάνελ να απαντήσουν. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Μπάρμπαρα Λοχμπίλερ είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα σχόλιο προς τον κύριο Γκαρσία. Εμείς, ένα περιφερειακό κοινοβούλιο, πρέπει να πω ότι ωφελούμαστε σημαντικά από τη δική σας δουλειά και ιδίω από το έργο που κάνατε εσείς ε, για την έννοια της ε, γυναικοκτονίας. Ήταν βάση της δικής μας δουλειάς. Άρα βλέπετε ότι βοηθά ένα τον άλλο. Και έχω και μια ερώτηση προς τον ε, καθηγητή Λούμπο. Το 2013 κάποιοι, εξημών και εγώ, πήγαμε στην Αφρικανική Ένωση και από ό,τι κατάλαβα, εκεί οι θεσμοί και οι μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι πολύ πιο μικροί σε σχέση με τις προσπάθειες που γίνονται για την πρόληψη των συγκρούσεων και την ερνευτική διαδικασία. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν για τις και που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Αντισαμπέμπα να έχουν πρόσβαση στους θεσμούς αυτούς ε, στα πλαίσια της Αφρικανικής Ένωσης. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι θα έλπιζα τουλάχιστον. Και επειδή έγινε μια συζήτηση σε σχέση με το Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο που εκπροσωπήθηκε στην προηγούμενη συνεδρία και υπάρχει από Αφρικανούς ηγέτες αρκετή κριτική που λένε πολύ αντί τα ε, εγκλήματα πολέμου και εγκληματίες πολέμου να διοκόντες σε αυτό το δικαστήριο καλό θα ήταν ε, να διευρυνθεί το έργο του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή η συζήτηση συνεχίζεται ή έχει σταματήσει καθότι έχουν, ξέρουμε, αποχωρήσει πολλά κράτη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λοχμπύρα, λέει ο πρόεδρος Λίβι Ολτιάν, Διεθνής Οργανισμός για την Πράσπιση των Θρησκευτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Εδώ είμαι. Α, εκεί πέρα είσαστε. Εκεί πίσω εξοχότητες και και κύριοι είμαστε αδελφιά ε, στην ανθρώπινη φύση αδέλφια συνάνθρωποι Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ σήμερα και εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΟΑΣΕ, το Συμβουλίο τη Ευρώπη, τα Ηνωμένα Έθνη και η οργάνωση που εκπροσωπώ. Το 1946 δημιουργήθηκε αυτή η οργάνωση και η κυρία Ρούσβελτ ήταν η πρώτη πρόεδρος. Εγώ εκπροσωπώ αυτή την, συνα... την οργάνωση σήμερα για τη θρησκευτική ελευθερία. Θέλουμε να εφαρμόσουμε την αρχή ε, αγάπη των πλησίων σε όσοι αυτός ή και παραπάνω. Έτσι θα έχουμε περισσότερη ειρήνη ασφάλεια. Κυρία Ρούσβελτ, από την αρχή, όταν ήταν η πρώτη πρόεδρος, υπό τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ εύκολα κατανοητά. Ελευθεροτύπη, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία του συνέρχεστε. Η ανάγκη να είναι κανείς ασφαλής στο σπίτι του. Να μην ε, τον ε, ε συλλαμβάνουν αυθαίρετα κτλ. Έχει να κάνει όχι μόνο με τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και με την κατεύθυνση προς την οποία οδεύουμε. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλω να τονίσω σήμερα. Από κοινού πρέπει να εστιάσουμε στην ελευθερία τη θρησκευτική, στην ελευθερία της σκέψης, του συνέρχεστε. Έτσι θα σεβαστούμε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα που δεν τη χάνουν επαρκώς προστασία στις κοινωνίες μας. Και έχω μια ερώτηση για τα μέλη του πάνελ. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε η ασφάλεια, η εθνική, η εθνική προστασία να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που να είναι σε βάρος των θρησκευτικών, εθνοτικών μειονοτήτων των προσφύγων και μεταναστών. Γιατί πολλές κυβερνήσεις σήμερα, όπως μια ανατολική, ανατολικοευρωπαϊκή χώρα, εκπονεί νομοθεσία που θα πλήξει τις θρησκευτικές μειονότητες. Πώς θα προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι καλύτερο για να προστατεύσει τι σχετικές ελευθερίες και αυτό το εκτιμώ, αλλά ε, θα ήθελα μια απάντηση. Ακίνα από το Παναφρικανικό Δίκτυο Πολιτών. Okay. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που με επιτρέπετε να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Η ερώτησή μου πάει στον Επίτροπο, στην Επίτροπο Λούμπου. Στην Αφρική πώς μπορούμε να εγγυηθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως για περιθωριοποιημένες κοινότητες όπως τους ΛΟΑΔ κατά πολιτικής αντιμετώπισης οι κυβερνήσεις θέλουν να αποφύγουν λογοδοσία τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν εξοπλίσει και προωθήσει το φόβο κατά μοαλοφιλοφίλων και καταπατούν τα δικαιώματα τους. Χώρες όπως η Ρουάντα και η Αίγυπτος έχουν κάνει επίθεση κατά της Επιτροπής και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ στην Αφρική. Χρησιμοποιούν τη φράση αφρικανικές αξίες σαν να ε, έτσι την απανθρωπιά και την ε, μυσαλλοδοξία να την στηρίζουμε μέσα από τις αφρικανικές αξίες. Ε, έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο στην Επιτροπή σαν πρόγραμμα υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά υπάρχει μεγάλη καταστολή και η παναχώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρε όπω είναι η Τανζανία. Έχουμε αυταρχικό καθεστώ και στρέφεται όχι μόνο κατά τον ΛΑΔ, αλλά και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Επίτροπε, ποιο ρόλο θα έχετε και εσεί και η Αφρικανική Επιτροπή όσον αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων, πώ θα αποκατασταθεί το ίχνος τη Αφρική για τα ανθρώπινα δικαιώματα πώς θα γίνει σεβαστή η αξιοπρέπεια όλων των Αφρικανών όπως βρίσκεται στη χάρτα την Αφρικανική Εθνοπίνων Δικαιωμάτων όπως και στην διακήρυξη που γιορτάζουμε σήμερα. Πιο συγκεκριμένα επίτροπο στατεύουμε την αξιοπρέπεια των ευάλωτων πληθυσμών της Αφρικής. Thank you, Madam Akina. And we have time for one more... Άλλη μια δήλωση ή ερώτηση. Έχουμε χρόνο. Ο Μαρ Φαρούκ από την Εθνική Ένωση των Δημοσιογράφων της Σομαλίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ο Μαρ Φαρού Κοσμάν, λέγομαι, είμαι από την Σομαλία και χαίρομαι όλους ιδιαίτερα που είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο. Διότι στη Σομαλία πολεμάμε. Μια κουλτούρα στη στιγματισμού και κατηγορίες κατά των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκείνων που κινούνται υπέρ τη ελευθερία έκφραση και υπέρ τη ελευθερία του συνεταιρία τη Σύμβατη Δημοσιογράφων. Και η χώρα μου είναι η πιο επικίνδυνη χώρα στην οποία μπορεί να είναι κανεί δημοσιογράφο στην Αφρική. Και χαίρομαι που ο Επίτροπο Ζερεμί ε, βρίσκεται στο πάνελ. Θέλω να δω τι συνεργασίε μπορούν να αναπτυχθούν κατά του στιγματισμού απονομιμοποίησης στα οποία υπόκεινται οι, πρόμα, οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική ε, και στη Λατινική Αμερική. Ρέμι και Ζωέλ, Πώ μπορείτε να συνεργαστείτε για να το καταπολεμήσετε αυτό και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υιοθέτησε ένα ψήφισμα περί τη καταστάσεω ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη Σομαλία 5 Ιουλίου φέτο. Αναφέρεται στο στιγματισμό των συνδικαλιστών, των δημοσιογράφων και εκείνων που πολεμούν για την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσαι στη χώρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στο τέλος που αναφερθήκατε στο σημαντικό ζήτημα που κάλυψε το Ευρωκοινοβούλιο στη Σομαλία. Στις 7 ακριβώ πρέπει να σταματήσουμε λόγω διερμηνίας. Έχουν δικαίωματα και αυτοί να τελειώσουν τη δουλειά τους. Δέκα λεπτά έχουμε. Κάθε μέλος του πάνελ θα έχει ακριβώς δύο λεπτά από την άποψή μου. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό, αλλά έτσι πρέπει να πράξουμε. Η ισορροπία των φίλων. Ξεκινήσαμε από τους άντρες. Να δώσουμε τώρα στα θηλυκά μέλη του πάνελ το λόγο πρώτα για να το εξορροπήσουμε αυτό. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, κύριε Ρούντολφ. Ευχαριστώ. Την ερώτηση Τη Ενώσεω για την προστασία των Σχετικών δικαιωμάτων, απαντήσω πρώτα. Θέσατε πολύ σοβαρό θέμα και πρόβλημα τη χρήση της εθνικής ασφάλειας σαν δικαιολογία για να περιοριστούν τα δικαιώματα των ανθρώπων. Όπως είπατε, δεν αφορά μόνο τις σκεφτικές μειονότητες, αλλά και άλλες μειονότητες, μετανάστες, επικριτές κυβερνήσεως κλπ. Δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση σε αυτό. Ο πλευράς των θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τι κάνουμε, ασκούμε τις διάφορες εξουσίες και δυνάμεις που έχουμε. Όταν συμβουλεύουμε τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, στηρίζουμε το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας. Δείχνουμε ότι είναι διακριτική μεταχείριση, έχει διακριτικές συνέπειες όταν αυτό συμβαίνει. Και ζητούμε να γίνει αξιολόγηση της νομοθεσίας και τι αντίκτυπο έχει μια νομοθεσία επί συγκεκριμένων ομάδων. Όπως έχουμε τη Γαλλική Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που το έκανε αυτό όταν υπήρχε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη Γαλλία για τους σκοπούς προστασίας εθνικής ασφάλειας και είχε διαφορετική, διαφορετικό αντίκτυπο για τις μειονότητες από ό,τι τους άλλους. Προσφεύγουμε και στα δικαστήρια. Προσφεύγουμε στα συνταγματικά δικαστήρια χωρών. Αυτή είναι η νομική πλευρά. Έχουμε και άλλη πλευρά. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία. Στην ανοιχτή συζήτηση να πηγαίνουμε εναντίον του αφηγήματος το αφηγήμα του χρησιμοποιούν οι διάφορες ομάδες. Θυμίζουμε στου πολίτε τι ευθύνε έχουν όσον αφορά το δημόσιο λόγο τους. Να μην προωθούν το ρατσισμό ή θρησκευτική διάκριση. Και μέσω εκπαίδευση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν λέμε απλώς τι είναι η νομοθεσία, τι αφορά η νομοθεσία, αλλά να αμεσω ποιες αξίες στηρίζουν τα ανθρώπινα νομοθεσια αλλα να καταλαβει ο κόσμο ποιε αξιες στηριζουν τα ανθρωπινα δικαιωματα και να υπάρχει και συνάντηση με εκπροσώπους των διαφόρων ε, κοινοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η κατανόηση περί Να καταλήξω σε κάτι που ήταν καθησυχαστικό. Η Γερμανία, σε Γερμανία 250 εκατομμύρια Άνθρωποι βγήκαν, διαδήλωσαν κάτω από το hashtag αδιέρετη. Είπαν ότι δεν πρέπει να είναι διχασμένη η κοινωνία, πρέπει να είμαστε μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητα ε, για το ποιο, ποια πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φροντίζουμε. Ευχαριστώ καθηγητά Ρούντολφ. Η κυρία Καταπαχάτσε έχει το λόγο. Θα σχολιάσω δύο πράγματα. Το πρώτο, ελευθερία της θρησκείας, η ανεξιθρησκεία και θέμα ασφαλείας. Έχουμε πονήσει ένα έγγραφο αυτό περιγράφουμε. Πού είναι τα σύνορα, η γραμμή διαχωριστική μεταξύ ασφαλεία και ανεξιθρησκεία. Πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια και πού ξεκινά η ανεξιθρησκεία και η ελευθερία τη θρησκεία που δεν πρέπει να υπονομευθεί εν ονόματι εθνική ασφαλείας. Το συζητούμε τι κυβερνήσει. Αυτό απαιτεί πολιτική βούληση βέβαια. Και έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Συνεργασία. έχουμε τεράστιο περιθώριο για βελτίωση. Για διεθνείς και περιφερειακούς μηχανισμούς. Μπορούν να μάθουν ένας από τον άλλον. Μπορούμε να διδάξουμε οι μεν τους δε. Μπορούμε να έχουμε συλλογική δράση. Όσο δρούμε μεμονωμένα, τότε η αποτελεσματικότητά μας είναι πολύ μικρότερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καθηγητά Πόμοντα, ακούσα αυτά που είπατε διότι μόλις επέστρεψα το πρωί από τον Καναδά, σήμερα. Να προσθέσω μια ερώτηση. Επικρίναμε την αντιμετώπιση των ηθαγενών πληθυσμών στον Καναδά. Άλλαξε η κυβέρνηση. Άλλαξαν τα πράγματα. Ή η κατάσταση είναι η ίδια όπως και επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Ευχαριστώ την ερώτησή σας. Είναι το πιο βασικό ερώτημα που με ερωτούν άνθρωποι από άλλες χώρες. Ήταν κατά των ηθαγενών ε, πληθυσμών η προηγούμενη κυβέρνηση. Ε, Θεωρούμεθα σαν απειλή κατά τη εθνική ασφάλεια. Και αυτό ο, ο Πρωθυπουργό λέει τα πάντα σωστά. Νύχτα με μέρα είναι η διαφορά. Ότι είναι σημαντική ε, θα κινηθούμε με βάση του ηθαγενεί του πληθυσμού που θέσουν τα δικαιώματα. Όλα επιδεινώθηκαν επί τη θητεία του. Να πω κάτι που απαντά και στο άλλο ερώτημα του άλλου κυρίου για την εθνική ασφάλεια και τον ευρύ αυτό φόσμο, το γενικό φόβο για το διεθνή ε, τρομοκρατία που υπονομεύει τι ατομικέ ελευθερίε στον Καναδά. Επί Πρωθυπουργού Χάρπερ πέρασε τον, τον νομοθεσία αντιτρομοκρατία που δεν αφορούσε καν τη διεθνή τρομοκρατία, αλλά αφορούσε οποιονδήποτε στον Καναδά που θα μπορούσε να παρέμβει στις διπλωματικές σχέσεις, στην οικονομία ή να επηρεάσει τις υποδομές. Και είχε συγκεκριμένο αντίκτυπο στοχευμένο επί των Ιθαγενών. Ανεξάρτητα από ε, όσα λέγονται, πάντα ειρηνικά διαδηλώναμε. Άοπλοι. Και θέλαμε φιλικά να βρούμε λύση. Αυτοί που πέθαναν στις διαμαρτυρίες ήταν μόνο οι δικοί μας τους σκότωσαν είτε οι αστυνομικοί είτε οι στρατιωτικοί. Θέλουμε να πούμε στου Καναδού ότι επιτρέποντα νομοθεσία αντιτρομοκρατική να είναι τόσο ολιστική, να καλύπτει τα πάντα και να απαρνείται τις θεμελιώδεις, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα των γενών είναι κάτι που μπορεί να καλύψει και εσά του λέμε. Και πρέπει όλοι μαζί να ανησυχούμε για αυτά. Και τελικά δεν τα καταφέρνουν μόνο τα λόγια, και το βλέπετε αυτό με τον τωρινό Πρωθυπουργό. Παρά το γεγονό ότι τα δικαστήρια λένε μην περάσουν από τα εδάφη των Ιθαγενών οι αγωγοί, έχουν συνταγματικά προστατευμένα δικαιώματα, λέει κοιτάξτε είναι τα συμφέρον τη χώρα, αυτό θα κάνουμε ούτω ή άλλω. Έχουν πραγματικό πρόβλημα στον Καναδά. Και άλλε χώρε θα πρέπει να το σημειώσουν αυτό, διότι αυτό επηρεάζει και τι διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε. Καλώ, ευχαριστώ. Καθηγητά απόμετρο, κυρία Γκαρθία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. σε ό,τι αφορά το σχόλιο της Λόχ Μπίλερ για το διαμερικανικό σύστημα και τις κτονίες φεμινισίδιο στην Ισπανία ή τις, τις λατινοαμερικανικές χώρες. Θέλω να αναφέρω κάτι για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη δουλειά μας. Συνεργασία κρατική. Οι διεθνείς οργανισμοί κάνουν ό,τι μπορούν. Και μπορούν να κάνουν πράγματα αν, έχουν, αν υπάρχει κρατική συνεργασία. Ουσιαστικά Είχαμε μια υπόθεση το 2009 κάπου Νέρο από τη Διαμερικανική Επιτροπή κατά του Μεξικού και συζητήθηκε στο Διαμερικανικό Δικαστήριο για την περίπτωση της επαρχής Τσιουάου ένα τζαμεκανό δικαστήριο απεφάνθη κατά του Μεξικού για τη διεθνή ευθύνη και για μέτρα ε, μη υποτροπής. Με αποτέλεσμα το Μεξικό υποχρεούται πλέον να, να εγκρίνει πολιτικές για να αποτραπούν οι δολοφονίες γυναικών και για να τιμωρηθούν οι δράστες. Το Μεξικό έχει προσυπογράψει την σύμβαση, έχει αναγνωρίσει την δικαιοδοσία του Διαμερικανικού Δικαστηρίου. Μέχρι στιγμής 20 μόνο αμερικανικά κράτη αναγνωρίζουν ε, τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου αυτού, άρα πολλά ακόμα απομένουν να γίνουν για να προωθήσουμε την προσχώρηση του, ε, στο δικαστήριο και την αναγνώριση αυτής ε, της προσπάθειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει, να προωθήσει δηλαδή ε, την προσχώρηση. Για τον Καναδά, για παράδειγμα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Δεν έχει προσπογράψει την Αμερικανική Σύμβαση ο Καναδά. Εξού και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διαμερικανικού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, Σα ευχαριστούμε κύριε Γκαρσία. Τέλο ε, ο καθηγητής Λούμπου. Γιατί και αυτός ε, έχει να απαντήσει κάποια προσωπικά ερωτήματα. Ναι, τρία τα ερωτήματα μέσα σε δύο λεπτά τι να πω και να πρωτοπώ. Καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέει ο πρόεδρο. Ναι, για το ότι δεν έχουν τι απαραίτητε δυνατότητε οι οργανισμοί και οι φορεί και τα λοιπά στον τομέα τη ασφάλεια και τη ειρήνη. Δεν ξέρω ποιο το ερώτημα, ε, αλλά θα έπρεπε να τα δει ε, πιο ανοιχτά τα πράγματα. Είναι πολιτικό το θέμα, δεν μένει στην Αντισαμπέμπα ούτε στο αφρικανικό ούτε στο διαμερικανικό ε, δικαστήριο. Το θέμα είναι να έρθει η ειρήνη και η δημοκρατία στην Αφρική. Για τις ΜΚΟ μπορούν να ζητήσουν καθεστώς παρατηρητή στην Αφρικανική Επιτροπή εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Και αν δεν τις πληρούν, ε, αποσύρεται αυτή η ιδιότητα. Αφαιρείται. Σε ό,τι αφορά το θεσπινικό ποινικό δικαστήριο. Αύριο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα δικαστήριο αυτή η ε, δικαιοδοσία που έχουμε τώρα, πολύ πιο ευρεία θα ε, είναι οι εξουσίε τη και ελπίζω να συμβεί σύντομα για το ΛΟΑΤ. Από τότε που ανέλαβα καθήκοντα, από τον Νοέμβριο δηλαδή, του προηγούμενου έτους, πάνω σε αυτό μόνο δουλεύει. Οι υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτοί που εργάζονται στον κλάδο αυτό, οι γυναίκε, οι υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ ή και ίδια άτομα αυτή τη κοινότητα αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλε δυσκολίε ακριβώ όλων των αφρικανικών αξιών. Ξέρω γιατί μιλάτε. Αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, οι αφρικανικέ αξίε δεν είδαν να είναι που ήταν εξ ονόματος αυτών νόμων, στο όνομα μάλλον αυτών, ξέρω τι υφίστανται οι ΛΟΑΔΜ. για τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων. Τα κράτη πρέπει να στήσουν να το κάνουν αυτό εγώ σε ένα συμπίλημα κάποιων αρχών για την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθώ να πάρω από όλου. Ε, τι κάνει το Συμβούλιο τη Ευρώ, Συμβούλιο τη Ευρώπη, ο ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν μπορούμε και εμεί στην Αφρική να ε, εμπνευστούμε. Όλα αυτά όμως είναι πολιτική, θέματα πολιτικής βούλησης και υπάρχουν δυσκολίες σοβαρές στην Αφρική. Και εμείς στις αποστολές προσπαθούμε να μιλήσουμε με τις κυβερνήσεις για να του πούμε ότι η περάσπιση των ανθρωπίνων δεν είναι έγκλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λούμπου. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Νομίζω Όπω ακούσαμε σήμερα, είναι σαφέ ότι είναι σημαντικό ο ρόλο των περιφερειακών ε, θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Για να αντιμετωπιστούν οι αλλαγέ ε, σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ και του οργανωτέ και σας καλώ, αν θέλετε, να χαλαρώσετε να δείτε την έκθεση για την Οικουμενική Διακήρυξη στο κτίριο Σπινέλ στον τρίτο όροφο. Σε λίγα λεπτά η Χάιντι Χάουταλα, αντιπρόεδρος, θα εγκαινιάσει στην έκθεση και θα ακούσετε και ένα μουσικό κονσέρτο στο Γεχούντι Μενουχίν, ε, στο Ισόγειο, στο ASP. Καλό βράδυ και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Έξω!